για παράδειγμα για τα μέταλλα έχω συζητήσει με, διά, διαφόρων κλάδων που λειτουργούν ε, με την ανοτεχνολογία ε, προσπαθούν να δημιουργήσουν εναλλακτικέ εκεί όπου οι σπάνιες γέες είναι δυσέβρετες Τέταρτη παρατήρηση είναι ανάπτυξη δικτών. Ζητώ από την Κομισιόν και τα κρατημέλη να επιταχύνουν τις διαδικασίες. Και πέμπτη προτεραιότητα είναι να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό. Αυτή τη στιγμή βασίζεται περισσότερο εστιάζει την προσοχή στην ενέργεια, αλλά θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο, κατά τη γνώμη μου, στο σχεδιασμό των προϊόντων και την δυνατότητα ανάκτησης υλικών που περιέχονται σε αυτά τα προϊόντα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στόχος για να μπορούν να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά οι πόροι. Αυτέ είναι οι πέντε δράσει προτεραιότητα. Φυσικά ήταν πολύ δύσκολο να περιοριστώ σε αυτέ τι πέντε προτεραιότητε, γιατί μπορώ να σκεφτώ ακόμα 10-20 άλλα πολύ σημαντικά ε, θέματα, αλλά κατέληξα σε αυτέ τι πέντε. Άλλα στοιχεία που θα βρείτε εδώ αφορούν τις κρατικές προμήθειες, αφορούν το ρόλο των καταναλωτών. Στο περσινό ευρωβαρόμετρο ε, φάνηκε ότι οι καταναλωτές είναι πρόθυμότατοι να συμμετέχουν ώστε να επιτευχθούν ψηλότερες προδιαγραφές ανακύκλωσης. Για παράδειγμα, πάνω από τα 3 τέταρτα των καταναλωτών είναι ενθουσιώδης και θα ήθελα να συμμετέχουν, να μετακινηθεί η φορολογία από την εργασία στην ρήπανση, ολόκληρο το θέμα των νέων μετρήσεων του ΑΕΠ μας και του πέρα από το ΑΕΠ, beyond GDP. Ο, περισσότεροι από αυτούς τους τομείς καλύπτονται σε αυτό το σχέδιο έκθεσης. Βέβαια, Έχω ακόμα τέσσερις σελίδες τροπολογίες για την ειδική μου έκθεση. Είναι αδύνατο να ανακαλυφθεί ένα τόσο ευρύ ζήτημα σε τέσσερις σελίδες. Θα τις δείτε την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω πως θα με βοηθήσετε να συμπληρώσω τα κενά που υπάρχουν στην έκθεση και προσβλέπω στις προτάσεις σας. Αλλά τέλος, και κλείνω έτσι πρόεδρε, θα ήθελα να σας καλέσω να προσπαθήσετε να μείνετε σε αυτό το σχεδιάγραμμα που σας έκανα, που σας παρουσίασα, να μείνουμε σε αυτές τις προτεραιότητες. Οι πέντε αυτές προτεραιότητες ίσως να μην είναι οι τελικές, αλλά ας προσπαθήσουμε να περιοριστούμε ώστε να έχει νόημα από πολιτική άποψη γιατί είναι πολύ σημαντικό απέναντι στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν κάτι τέτοιο και ελπίζω πως θα μπορέσετε να συμφωνήσετε μαζί μου. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Κερπλάντη. Προχωράμε τώρα στην συζήτηση με τους κοιόδες εισηγητές. Πρώτα ο Καρλ Χάιτς Φλόρενς, μετά η Ιούντιθ Μέρκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, αγαπητέ συνάδελφε κύριε Κερπράντη, ε, μας έχετε υποβάλει την έκθεσή σας. Ε, έχουμε... Είχαμε την ευκαιρία να έχουμε κάποιες συζητήσεις. Συμφωνώ με το ότι έχετε εγκαταλείψει τον πολύ αυστηρό δρόμο που υπέδειξε η και που ε, συμβάλλεται εδώ με νέα στοιχεία και αναφέρεται μια νέα οπτική των πραγμάτων. Αυτό το βρίσκω πολύ θετικό. Θα ήθελα ρητά να στηρίξω ε, αυτό που είπατε ότι δεν σας ενδιαφέρει να έχουμε τόσες πολλές ε, τροπολογίες. Δεν θέλουμε να ε, διακυβεύσουμε την όλη διαδικασία. Σίγουρα υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία θα θέλαμε να τονίσουμε. Ε, συμμερίζομαι τους ε, τομείς κλειδιά. Ε, θα πρέπει να προωθηθεί η αγορά των δευτερευόντων υλικών Πιστεύω επίση ότι είναι πολύ καλή η προσέγγιση σας ε, που αφορά ε, τον τομέα Schengen. Ε, θα πρέπει να κοιτάξουμε και το θέμα των φόρων και αυτό συνδέεται με το θέμα αυτό. Πιστεύουμε ότι αν με τους φόρους μπορούμε να καθοδηγήσουμε τις τάσεις, αυτό είναι καλό και θα πρέπει να το συζητήσουμε. Εμένα με προβληματίζει ο οικολογικός σχεδιασμός. Και το ότι στον τελικό λογαριασμό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει κανείς και το κόστος του οικολογικού σχεδιασμού. Ο γιος μου καλλιεργεί δέντρα. Εάν σε ένα εκτάριο έχει καλλιεργήσει 500 δέντρα, Ε, και τα πουλήσει αυτά, τότε τι είδους οικολογικό σχεδιασμό θα συμπεριλάβει στο λογαριασμό. Είναι σαφής για μένα ο βασικός ορισμός του οικολογικού σχεδιασμού, αλλά νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε πώς θα χειριστούμε το θέμα αυτό. θα πρέπει ε, να φροντίσουμε να χειριστούμε το θέμα αυτό σωστά για να μην πλέξουμε σε ατελείωτες διαδικασίες. Όσον αφορά τους δείκτες σας, και εγώ είμαι υπέρ των ε, δικτών, αλλά νομίζω θα προτιμούσα έναν ανοιχτό κατάλογο. Δεν είμαι βέβαιος αν γνωρίζουμε ακριβώς γιατί οι δείκτες μιλάμε και πόσο θέλουμε να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό. Θα ήθελα και σε αυτόν τον τομέα μια διευκρίνηση ε, από την μελέτη επιπτώσεων. Θα ήθελα επίσης ε, να αναφερθώ στο θέμα των ε, φόρων. Νομίζω ότι είναι σωστό αυτό που είπε η κυρία Χέντεγκάρτ ότι θα πρέπει να, ε, ε, να φορολογούμε αυτά που καταναλώνουμε, όχι αυτά που παράγουμε. Αλλά θα πρέπει να αλλάξει η φορολογική ε, πολιτική στην Ευρώπη. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Θα πρέπει να ακούσουμε και τα επιχειρήματα αυτών που λένε ότι θέλετε να φορολογήσετε την κατανάλωση, δεν θέλετε να μειωθεί όμως ε, αλλά δεν θα, δεν θα μειώσετε αλλού την φορολογία. Ε, βλέπω ότι αυξάνεται στη χώρα μου η φορολογία σε κάποιου τομεί, ε, δεν μειώνεται σε άλλου ε, τομείς. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί. Ωστόσο, θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα και πολύ ε, ε, ευχαρίστως ε, θα στηρίξω το θέμα αυτό με μετριοπάθεια. Ε, οι συνάδελφοι που έχουν αποφασίσει να γίνουν χορτοφάγοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ε, το αποτέλεσμα που θα πετύχουν σε σχέση με, τους, με αυτούς που τρώνε κρέας ε, θα είναι σαν να μειώσουν την ε, θερμοκρασία στο σπίτι τους για τρία άτομα από 23 σε 22 βαθμούς. Μην νομίζετε λοιπόν ότι μπορείτε να σώσετε τον κόσμο αν δεν τρώτε κρέας, αλλά βέβαια ο καθένας σας το κάνει όπως θέλει. και θα πρέπει ε, να κοιτάξουμε και ε, ε, και την ορολογία που χρησιμοποιούμε εδώ, διότι μιλάμε για απόβλητα. Αυτό είναι κάτι αρνητικό. Η ανακύκλωση Είναι και αυτή ένα θέμα. Βλέπω στην... Ε, βλέπω στη χώρα μου ότι ο κόσμος ε, ε, συλλέγει σαν τρελός τα ανακυκλώσιμα, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να τα ανακυκλώσουμε σωστά. Δηλαδή χωρίζουμε τα άσπρα από τα καφέ μπουκάλια, αλλά τελικά έρχεται το φορτηγό και τα ανακατεύει μεταξύ τους. Νομίζω θα πρέπει να προχωρήσουμε με περισσότερη ακρίβεια στον τομέα αυτό και να δούμε ποια είναι τα συγκεκριμένα βήματά μας ε, στην ε, διαδικασία της ανακύκλωσης, ε, ώστε να μπορούμε να έχουμε πρότυπα. Κατά τα άλλα, συνάδελφε Κερβράντη, θα χαρώ πολύ να συνεργαστώ μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φλόρενς η ε, σκιώδη συγγήτρια Γιούντιθ ε, ε, Μέρκης και κατόπιν ο Άικχαουτ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον συνάδελφο για την ε, εξαιρετική του παρουσίαση και έκθεση. Και σας ευχαριστώ πάνω απ' όλα για το ότι εστιαστήκατε στην καινοτομία. Συμφωνώ μαζί σας. Βέβαια θα πρέπει να διευκρινίσουμε τι είδους καινοτομία εννοούμε. Και έχω κάποιες ιδέες. Very Θα πρέπει να αποφύγουμε ενοχλητική καινοτομία. Δηλαδή, ο υπολογιστής άλλαξε τον κόσμο μας. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα, δεν ξέρω, δημοσιονομικό, τεχνικό. Πάντως θα πρέπει κάπως να αλλάξουμε τον τρόπο που προσεγγίζουμε τους πόρους. Attention, therefore, on the, reference. Αναφερθήκατε στην Ένωση της Καινοτομίας. Πολύ σημαντική μνήμα αυτή και ε, καλό είναι να συνδεθεί και με τη στρατηγική για τις πρώτες ύλε που εγκαινιάστηκε πέρυσι. Έχαμε συντάξει και σχετική έκθεση. Και τότε είχαμε καταλήξει σε κάποιες κοινέ θέσει που θα ήθελα να επαναλάβω και σήμερα. Σε ό,τι αφορά την πρότασή σας, για μια δημοσιονομική αλλαγή, φορολογική αλλαγή. Συμφωνώ, αλλά είναι κάπως αόριστη, απροσδιόριστη η πρότασή σας. Γιατί λέτε να γίνει μια μεταστροφή του βάρους μεταξύ της φορολογικής, περιβαλλοντικής φορολογίας και των εισοδημάτων. Βέβαια, αν προσθέσετε κάτι, όπως είπε ο κύριος Λόρες, θα πρέπει να αφαιρέσετε κάτι. Και είπατε μετακίνηση, δηλαδή μετατόπιση από κάτι σε κάτι άλλο. Πού έγινε η μετατόπιση από την εργασία, όπως είπατε, από την επιβάρηση της εργασίας σε ε, φορολογία πρώτων υλών. Πραγματικά χρειαζόμαστε μια ισχυρή φορολογική βάση, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το φορολογικό μας σύστημα για να δώσουμε κίνητρα και για τα προγράμματά μας για την αξιοποίηση των πόρων και κάπου θα πρέπει να προσδιορίσουμε και να συγκεκριμενοποιήσουμε το θέμα αυτό. Συμφωνώ απόλυτα και με τον κύριο Κερπράντη και με τον κύριο Φλόρενς ότι με το φορολογικό μας σύστημα θα μεταρρυθμίσουμε και την κοινωνία. Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο στο φορολογικά ζητήματα και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Κάτι άλλο που λείπει δυστυχώς από την έκθεση είναι πώς θα αποφύγουμε ένα είδος μπούμεραν. Γιατί αν είμαστε αποτελεσματικοί πώς θα αποφύγουμε το να γίνουν όλο και πιο φθηνά τα προϊόντα και άρα να αυξηθεί η κατανάλωση. Προσοχή να μην έχουμε αντίθετα αυτά τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Κάτι άλλο που φαντάζομαι θα σας ε, απασχολεί ήδη είναι ότι ο κινητήριος μοχλός της κοινωνίας είναι είτε μια αλλαγή της ε, καταναλωτικής συμπεριφοράς, είτε ε, μια αλλαγή στο επιχειρηματικό μοντέλο, είτε ένα συνδυασμό των δύο. Υπάρχουν διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα, οπότε καλό θα ήταν να ενθαρρύνουμε τον ιδιωτικό τομέα να αναθεωρήσει τα επιχειρηματικά μοντέλα και θα μπορούσαμε και εκεί εμείς να δώσουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Ε, δεν ξέρω αν θα πρέπει να έχουμε μια κοινωνία περι, περισσότερο μίσθωσης παρά α, κυριότητας των προϊόντων. Να προωθήσουμε δηλαδή την ανακύκλωση αντί για την κυριότητα, την ιδιοκτησία των προϊόντων, να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ε, ε, μίσθωση, στην προσωρινή κατοχή. Τώρα, για τα απόβλητα, διαχείριση απόβλητων πολύ σημαντικό. Θα πρέπει ε, να έχουμε μία ιεράρχηση των αποβλήτων, μία ε, ιεράρχηση των ε, πρώτων υλών και των πόρων μας. Να χρησιμοποιούμε, να αξιοποιούμε στο έπακρο τις πρώτες ύλες μας. Όπως είπατε ότι ίσως δεν είναι σε εμά να καθορίσουμε την ιεραρχία, την ιεράρχηση αυτή των πρώτων υλών, αλλά θα μπορούσαμε τουλάχιστον να δώσουμε τον αρκτήριο λάκτισμα στη συζήτηση κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να επαναφέρουμε στη συζήτηση είναι ότι έχουμε ένα ποσοστό, ένα συντελεστή συγκέντρωσης για τα απόβλητα, αλλά δεν είναι ε, το, ο βασικός μας στόχος για τα δευτερογενή υλικά. Αναφέρθηκαν ε, κάποια υλικά ε, όπως ε, χρυσός ή θείο, αλλά Σίγουρα εδώ η εμπειρογνωμοσύνη, η τεχνογνωσία είναι σημαντική. Δεν μα ενδιαφέρει μόνο ο συντελέστή συγκέντρωση του θείου, αλλά και ο συντελεστή συγκέντρωση των πολύτιμων λίθων, των πολύτιμων υλικών. Σε ό,τι αφορά τα δευτερογενή προϊόντα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φυσικά τη φορολογία, όπω είπατε, αλλά όπω είπατε και εσεί, πολλοί κανόνε μα εμποδίζουν να χρησιμοποιήσουμε δευτερογενή υλικά. Υγειονομικοί κανόνε, για παράδειγμα οι κανόνες υγείας, υγιεινής. Χρειαζόμαστε μια ισορροπία, γιατί θα, πρέπει να θεωρούμε τους κανόνες μας για να εξακριβώνουμε κατά πόσο είναι αποτελεσματική σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των πόρων. Να δοκιμάζουμε τους κανόνες μας συνέχεια και να δούμε αν είναι σωστοί. Δώσατε μεγάλη έμφαση στον ιδιωτικό κλάδο σε ό,τι φορά το καταναλωτή, αλλά νομίζω ότι δεν θα πρέπει να ξεχνούμε και τον καταναλωτή. Ναι, μεν ε, εστίαση στον ιδιωτικό κλάδο, αλλά να μην ξεχνάμε και τον καταναλωτή. Το θέμα της διατροφής πολύ σημαντικό να αναφέρεται στην ε, έκθεση, ότι καλό θα ήταν να αλλάξουμε τον τρόπο διατροφής μας. Αυτό θα επηρεάσει και τον τομέα των μεταφορών αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να, τρο... να αλλάξουμε την καταναλωτική μας συμπεριφορά, όχι μόνο τη διατροφή μας. Ας μην ξεχνούμε λοιπόν όχι μόνο την, ε, ε, και την ευθύνη του καταναλωτή, γιατί μιλάμε για την ευθύνη του παραγωγού, αλλά και ο καταναλωτής έχει κάποια ευθύνη. Και να δούμε και τις ετικέτες, τη σήμανση που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να έχουμε μια ολοκληρωμένη ετικέτα που να αναφέρει και το fair trade, το δικαιομπόριο, την ε, ενεργειακή αποδοτικότητα, να δίνει πολλές πληροφορίες στον καταναλωτή για την προέλευση, τη χρήση και την, τον τελικό προορισμό ε, του προϊόντος και γενικώ πληροφορίες για όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος δεν είμαι και πολύ ενθουσιώδης ε, για την ανατεχνολογία, τα ανανοηλικά. Δεν συμμερίζομαι τουλάχιστον το δικό σας ενθουσιασμό, γιατί μερικές ε, ε, ε συνέπειες των ανανοηλικών ε, είναι ακόμη απρόβλεπτες. κοιτάξτε τι συμβαίνει με τον άργυρο. Ε, πολλές φορές μπορούν να αποβούν εις βάρος της βιοποικιλότητας ο τρόπος ε, ε, αποσύνθεσης αυτών των ανανοηλικών. Ως προς τα απόβλητα. Καλό θα να χρησιμοποιήσουμε τα απόβλητα και να τα αξιοποιούμε, αξιοποιούμε τη διαχείριση του στο έπακρο. Αλλά για το Σέγγεν δεν είμαι σίγουρη. Δεν πρόκειται να κατονομάσω χώρες βέβαια. Αλλά κάποιες χώρες στην Ευρώπη δεν έχουν τόσο καλές επιδόσεις όσο οι υπόλοιπες. Οπότε έχουμε πολύ καλές νομοθετικές διατάξεις ε, για τη ε, διαχείριση αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν εφαρμόζονται πάντοτε. Από τη στιγμή λοιπόν που οι κανόνες μας δεν εφαρμόζονται αποτελεσματικά, εγώ είμαι κατά της πρότασης χώρου Σέγγεν γι' αυτό. Γιατί ε, αυτό που χωλαίνει στην όλη κατάσταση είναι η εφαρμογή, όχι η νομοθεσία. Αυτά και ελπίζω να βελτιώσουμε με την περαιτέρω συζήτηση και τις τροπολογίες και την έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Ιούτιτ Μέρκης. Ε, ο Πας παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον ε, Ιαν για την έκθεση του που πραγματικά προσδιορίζει ένα πολύ σωστό πρόγραμμα για το θέμα αυτό και μπορώ να σας διαβεβαιώσω για την υποστήριξη, τη θερμή υποστήριξη των πρασίνων γιατί και εμεί ε, θέλουμε αυτό το πρόγραμμα να αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό τη οικονομία στην Ευρώπη στο μέλλον. Και ευελπιστούμε ότι η έκθεση αυτή θα προκαλέσει ε, ευρεία συζήτηση, όχι μόνο στη δική μα Επιτροπή, την Επιτροπή Περιβάλλοντος, αλλά και σε άλλε επιτροπέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί εκεί έγινε το πρόβλημα. Το χρησιμοποιούμε όταν μιλούμε για αξιοποίηση των πόρων. Θεωρούν πολλοί ότι είναι θέμα που αφορά μόνο το περιβάλλον, την Επιτροπή περιβάλλοντο. Λάθο είναι κατεξοχήν οικονομικό το πρόγραμμα, γιατί αυτό θα αποτελέσει το κινητήριο μοχλό της Ένωσης, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ζωτική σημασία σε αυτό το θέμα και δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Δεν αφορά μόνο τις περιβαλλοντικές ανησυχίες. Θέλουμε να διευρυνθεί η συζήτηση, να ξεπεράσει τα όρια, τα στενά όρια της δικής μας Επιτροπής και θα σας βοηθήσουμε. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή αφετηρία η έκθεσή σας. Όπως είπατε και εσείς όμως, Ήδη έχετε καταρτήσει και στις τροπολογίες και εμείς το ίδιο. Και θα ήθελα να επικεντρωθώ εδώ σε τέσσερα σημεία. Το θέμα του mainstreaming, το θέμα των αποβλήτων, της τιμολόγησης και το επίπεδο φιλοδοξιών της ε, έκθεσής σας. Σε αυτά τα τέσσερα σημεία ελπίζω να συμβάλλουμε για να ενισχυθεί η έκθεση και φυσικά παραλαμβάνω να επεκταθεί η συζήτηση και εκτός Επιτροπής. Ας ξεκινήσουμε με το mainstreaming. Καταρχήν, σας καθησυχάζω, δεν πρόκειται να τροποποιήσουμε τη δομή της έκθεσής σας, επουδενή. Θα ήθελαμε κι εμείς μια ιεράρχηση. Δεν θέλουμε ε, να προσθέσουμε ένα κατάλογο, ένα ευχολόγιο ε, πέραν των δικών σας προτεραιοτήτων, γιατί νομίζω ότι καλό θα ήταν να διαφυλαχθεί η δομή της έκθεσης, να βελτιωθεί φυσικά, να γίνει πιο οξυδερκής, πιο ισχυρή. Τώρα, ως προς το mainstreaming. Εμείς ε, θα θέλαμε φυσικά να συμπεριληφθεί αυτό το πρόγραμμα στη στρατηγική του 2020 και να καταλήγει σε βασικούς δείκτες που θα ληφθούν υπόψη στη μελλοντική οικονομία. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι στην Ευρώπη μας ενδιαφέρει η δημοσιονομική εξυγίαση, σίγουρα, αλλά σε τελική ανάλυση, αν δεν προσαρμόσουμε την οικονομία μας προς, την, προς το στόχο της αξιοποίησης των πόρων, θα, θα εξακολουθήσουμε να έχουμε προβλήματα με τους προπολογισμού, γιατί θα είναι ε, υπερβολικά δαπανηροί οι πόροι μας. Οπότε Αναφέρεται και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική του 2020, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, αλλά θα θέλαμε μια πιο κατηγορηματική διατύπωση ό,τι αφορά την παραγωγή και την κατανάλωση. Θα πρέπει να τονίσουμε και αυτού του κρίκους τη αλυσίδα, τη παραγωγή και τη κατανάλωση. Και σε ό,τι αφορά τη φορολογική μεταρρύθμιση, και εκεί θα σα βοηθήσουμε. Τώρα, για τα απόβλητα, το δεύτερο σημείο. Συμφωνώ με τη Γιούδιθ. Και έχω κι εγώ επιφυλάξεις για την πρότασή σας ε, για το Σέγγεν. Καλή ιδέα για ζώνη Σέγγεν, εφόσον έχουμε μια ιεράρχηση των αποβλήτων. Από τη στιγμή όμως που δεν έχουμε, ας μην ξεκινήσουμε ανάποδα. Από τη στιγμή που δεν έχουμε ιεράρχηση των αποβλήτων, δεν έχει νόημα το Σέγγεν. Πολλό δε μάλλον που πολλές χώρες δεν πληρούν καν τις προποθέσει δεν εφαρμόζουν καν τους κανόνες που ήδη υπάρχουν. Πρώτα χρειαζόμαστε μια ιεράρχηση των αποβλήτων και κατόπιν να φτάσουμε σε ένα σχεδόν μηδενικό υπόλοιπο αποβλήτων. Δηλαδή μετά την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση να μην μας μένουν καν απόβλητα. Πρώτα σε αυτό το σημείο να δώσουμε έμφαση και μετά να ξεκινήσουμε με την ιδέα της Schengen West. Πολύ προσοχή λοιπόν, γιατί να μην ξεκινήσουμε να εξομοιώνουμε τη μεταφορά αποβλήτων με τη μεταφορά ειδωτός. Είναι πολύ αναποτελεσματικό κάτι τέτοιο. Η γενική δεν μπορεί να είναι καλή, αλλά όχι προθύστερο σχήμα. Πρώτα η ιεράρχηση αποβλήτων και μετά συζήτηση για τη ζώνη Σέγγεν ως προς τα απόβλητα. Κάτι άλλο που λείπει από την έκθεση είναι μια ε, επίκριση εκεί που είμαστε ε, συνεπείς στην έκθεση για, τα ανανεώσιμα, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προ, προτείνουμε αναποτελεσματικούς τρόπους για, τις, για τα εργοστάσια που χρησιμοποιούν ε, άνθρακα. Γιατί μερικές, είπαμε να χρησιμοποιούμε τη βιομάζα για ενέργεια, αλλά όχι να την καίμε με ένα αποτελεσματικό τρόπο δεν είναι αποτελεσματική η χρήση της βιομάζας που προτείνεται στην οδηγία για τα ανανεώσιμα. Προσοχή λοιπόν στην ιεράρχηση. Ω προ το σημείο αυτό χρειάζεται κάποια ενίσχυση της έκθεσης. Θα σας βοηθήσουν οι πράσινοι, γιατί φαντάζομαι ότι και οι δικέ σας αυτό το στόχο θα έχουν, αλλά και οι δικές μας το ίδιο. Σε ό,τι αφορά την τιμολόγηση. Και ω προς το σημείο αυτό η έκθεση χρήζει κάποια ε, ενίσχυσης. Νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει κατεξοχήν να αναγνωρίσουμε είναι ότι αν δούμε πώς ε, βελτιώσαμε την ε, παραγωγικότητα ε, της εργασίας σε σχέση με την παραγωγικότητα των πόρων, διαπιστώνουμε που έγινε το πρόβλημα. Στις τιμές ανέκαθεν επιβάλαμε φόρο στην εργασία, κάτι που οδήγησε σε μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, που είναι θετικό μεν, αλλά αν κοιτάξουμε την ε, από παραγωγικότητα των πόρων, την αποδοτικότητα των πόρων, βλέπουμε ότι αυτή μειώνεται. Και αυτό ε, οφειλόταν στην επιβολή του βάρους της τιμολόγησης. Γιατί σε τελική ανάλυση έτσι θα αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των πόρων. Και εκεί θα σας βοηθήσουμε. Τέταρτο και τελευταίο σημείο, το επίπεδο της φιλοδοξίας της έκθεσης. Σε ορισμένα σημεία νομίζω θα μπορούσαμε να είμαστε πιο απαιτητικοί. Λέτε, ενθαρρύνουμε ή απευθύνουμε έκκληση για δράση. Όχι. Θα πρέπει να είμαστε πιο σαφείς. Για τα ορόσημα. Είπατε ότι ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε στόχους. Αλλά και εκεί μπορούμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Μιλήσαμε για αποσύνδεση της οικονομικής μεγέθυνσης. Να μιλούμε για παντελή αποσύνδεση της οικονομικής ε, μεγέθυνσης. Και εκεί λοιπόν πιο φιλόδοξη σε ό,τι αφορά τους δείκτες. Ναι, να έχουμε δείκτη παραγωγικότητας των πόρων, αλλά αυτό έχει περισσότερο επικοινωνιακό σκοπό. Αλλά τι γίνεται με το ε, αποτύπωμα γης, ύδατος και άνθρακα. Γιατί ωραία ακούγεται για κάποια περιοδικά ο δείκτης ε, παραγωγικότητας πόρων, αλλά στην ουσία είναι κάπως ασαφές να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Σίγουρα θα υποβάλουμε πληθώρα τροπολογιών και ως προς αυτό το σημείο. Πάντως, γενικά υποστηρίζουμε την έκθεση, θα την ενισχύσουμε και θα την επεκτείνουμε πέραν της Επιτροπής Περιβάλλοντος, γιατί από αυτή εξαρτάται το μέλλον της οικονομίας μας. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής είναι ο Μύρος Ναυσρούσκη, σχεδόν συζητητής για το ECR. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να συμφωνήσω με τους συναδέλφους που ευχαρίστησαν τον κύριο Γερμπράντη για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει. Μου αρέσει πολύ η δομή της έκθεσης ε, και σίγουρα θα στηρίξω τον καθορισμό προτεραιοτήτων στην Ευρώπη. Είμαι βέβαιος ότι θα είναι εύκολο να συντάξουμε, ότι θα είναι δύσκολο να συντάξουμε έναν κατάλογο ε, επιθυμιών. Συμφωνώ όμως με τον κύριο Γερμπράντη ότι ε, είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε ε, σε λίγα σημαντικά θέματα τα οποία θα αποτελούν το αποτέλεσμα συμβιβασμού. Βρίσκω θετική και την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην όλη διαδικασία. Έχω επικρίνει στο παρελθόν κάποιες προτάσεις της Επιτροπής μας, βρίσκω όμως την ε, ενεργειακή απόδοση ζωτική σημασία για την Ευρώπη, όπως άλλωστε και για τον υπόλοιπο κόσμο. Και πιστεύω ότι η πολιτική μας θα πρέπει να αποτελέσει κίνητρο. Συμφωνώ και με την ανακύκλωση υλικών. Και στις περιπτώσεις όπου είναι αδύνατη η ε, ανακύκλωση, να χρησιμοποιούμε τα απόβλητα για την ε, παραγωγή ενέργειας. Συμφωνώ με την ιδέα ότι η διαχείριση των αποβλήτων ε, θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο τοπικών αποφάσεων. Εάν κάποιος που μένει κοντά στα σύνορα της Τσεχίας δεν έχει αντίρρηση να εισάγονται ε, απόβλητα από την Γερμανία, δεν καταλαβαίνω γιατί να απαγορεύσει την πρακτική αυτή το Ευρωπαϊκό Βουλίο. Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι πριν 10 χρόνια ε, κάποιες χώρες ε, της ε, Δυτικής Ευρώπης διέθεταν τα αποβλητά τους πουλώντας τα φτηνά σε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Και έτσι δημιουργήθηκαν παράνομες χωματερές και στη χώρα μου και... Ήδη σήμερα προσπαθούμε να διαχειριστούμε τα απόβλητα αυτά, θα χρειάζεται προσοχή. Πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί όσον αφορά τα κριτήρια παραγωγής. Είναι δύσκολο να αποφασίσει κανείς σε κεντρικό επίπεδο τα βήματα που θα πρέπει να ληφθούν για την ενεργειακή απόδοση. Φοβάμαι ότι κάποια γραφειοκρατικά μέτρα και βήματα μπορεί να ε, δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα ε, παρά όφελος. Έγινε μια μακρά συζήτηση για την απαγόρευση των ε, κλασικών γλόμπων θέλαμε να μειώσουμε τη χρήση ε, ε, ε, υδράργυρου στα, στους γλόμπους και με ρώτησαν γιατί δεν απαγορεύουμε τα... Γιατί απαγορεύουμε τη χρήση των κλασικών θερμόμετρων, επιτρέπουμε όμως την χρήση υδράργυρου σε ακριβούς γλόμπους υψηλής κατανάλωσης που ε, ε, δεν είναι και καλή για την υγεία των ανθρώπων. Ε, θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τη θέσπιση κριτηρίων για τα διάφορα προϊόντα. Θα ήμουν επίσης ε, ιδιαίτερα επιφυλακτικός όσον αφορά οποιαδήποτε πτυχή συνδέεται με τη φορολογία. Πιστεύω ότι η φορολογία είναι κάτι που εμπίπτει απολύτως στην αρμοδιότητα των κυρίαρχων κρατών μελών και οποιαδήποτε προσπάθεια από πλευρά μα ή από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσουμε πανευρωπαϊκό σύστημα φορολογία. Θα έβρισκε την πολιτική μου ομάδα αντίθετη. Κατά τα άλλα, πάντως, ε, σας ευχαριστώ για την ε, εξαιρετική έκθεσή σας. Θα είναι ε, χαρά μας να συμβάλλουμε στη διαμόρφωσή της στο μέλλον. Έτσι ολοκληρώσαμε τον κύκλο των σκιωδών εισηγητών και διαβάζω τον κατάλογο των επόμενων ομιλητών. Και κλείνω τον κατάλογο των ομιλητών. Έχουν στήσει το λόγο. Dann Frau dann Herr Couchet, Herr Schnellhardt, Satuhassi, Richard Seber und Adam Gierig. Yes, you're, you're the first one. Äh, ich würde vorschlagen, damit der Zeit... Äh, Jana, ε, μην ξεφύγουμε από το χρονοδιάγραμμα και να μπορέσει να απαντήσει και ο εισηγητής σε ερωτήσεις και να πάρει το λόγο και η Κομισιόν να περιοριστούμε στα δύο λεπτά, ώστε να μπορέσουν όλοι να θέσουν τις ερωτήσεις τους. Από ό,τι βλέπω ε, συμφωνείτε. Προχωράμε λοιπόν. Η συνάδελφος Χίμνερ έχει πρώτο λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι ειλικρινά και Συγχαίρω τον συνάδελφο για τη θέση που έλαβε και για την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Γιατί αν θέλουμε να προσθέσουμε πολλά και διάφορα θέματα, θα αποσπαστεί η προσοχή μας από τα πιο σημαντικά. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά τους πόρους μας. Βέβαια γίνεται μια διάκριση ε, των πόρων, ανάλογα με την προέλευσή τους, αυτών των υπαρχόντων, των πρώτων υλών δηλαδή, που θα εξοριχθούν, που ήδη υπάρχουν ή που θα ανακαλυφθούν, θα, τους αναζητήσουμε σε νέες, θα τις αναζητήσουμε σε νέες πηγές, αλλά θα πρέπει να ε, χρησιμοποιήσουμε εκτεταμένα την ανακύκλωση, ιδιαίτερα των σπάνιων ε, υλικών, των σπάνιων ε, μετάλλων, που χρειάζονται ιδιαίτερα στην ηλεκτρονική και ηλεκτροτεχνική. Επίσης, τι γίνεται με τις χωματερές που λειτουργούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ίσως ε, και από εκεί θα μπορούσαμε να αντιλήσουμε κάποια υλικά, κάποιες πρώτες ύλες. Ε, στους χώρους ταφής, συγγνώμη, όχι στις χωματερές, στους χώρους ταφής μπορεί από εκεί να αντιλήσουμε κάποια υλικά. Τα δάση μας είναι φυσική πηγή βιομάζας ε, που χρησιμοποιείται μερικές φορές ε, κατεξοχήν αντί να αναδασώνουμε όλο και περισσότερο. Και μην ξεχνάμε στους σπόρους μας και το είδωρ που μπορεί να ε, αξιοποιηθεί πολύ αποτελεσματικά. Ή επίσης ε, ο άνεμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Θα πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε τους σπόρους μας και ας μην ξεχνάμε αυτά που μας είπε ο κύριος Φλόρεντς. Μιλάμε για αξιοποίηση των απορριμμάτων αλλά όταν μιλούμε για απόρριμα σημαίνει ότι ήδη δεν χρησιμοποιείται πια γιατί πηγαίνει στη χωματερή. Λέμε ότι ε, το απόρριμα μιας ε, βιομηχανίας μπορεί να αποτελέσει πρώτη ύλη για άλλη βιομηχανία. Μην το ξεχνούμε και αυτό. Δεν είναι όλα απόβλητα. Η επιτήρηση, το monitoring θα πρέπει να γίνει σε διακρατικό επίπεδο, να αναζητήσουμε καινοτόμε λύσει και σε ό,τι αφορά τις φορολογικέ προτάσεις ή του φόρου ε, θα πρέπει στόχο να έχει φορολογία τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και την προαγωγή της καινοτομίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Συγκητά πιστεύω ότι αυτό το σχέδιο έκθεσης του ψηφίσματος είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και οι συνάδελφοι ήδη ανέφεραν τις διάφορα, τα, τα διάφορα πλανεκτήματά του. Θα ήθελα ωστόσο να διευκρινίσω κάποια πράγματα και να σας θέσω ερωτήσεις κύριε Σιγητά. Μετά λέτε για καλύτερη χρήση των πόρων. Αν θέλουμε όμως να είμαστε λίγο πιο λεπτολόγοι σε αυτή την ε, λέξη πόρους θα έπρεπε ίσως να διακρίνουμε τους ανανεώσιμους από αυτούς που δεν είναι ανανεώσιμοι και έπειτα υπάρχει και μια διάμεση κατηγορία πολύ μεγάλη που είναι οι ανακυκλώσιμοι πόροι που απαντώνται και στα δύο ήδη, ανανεώσιμος και μη ανανεώσιμος. Το ίδιο, το ίδιο συμβαίνει με το νερό. Το νερό είναι ανακυκλώσιμο. Το ίδιο νερό έχουμε στη γη εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια, αλλά πρέπει να δούμε αν είναι μολυσμένο ή όχι κτλ. Μήπω θα ήταν λοιπόν πιο λεπτό και πιο αποτελεσματικό τουλάχιστον να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στου ανακυκλώσιμου και μη πόρου. μιλάμε για στερεά καύσιμα στερεά ε, που βρέχεται από ρηκτά ε, καύσιμα ή πρωτεσίλες όπως κάποια μέταλλα και τις ε, πόρους που είναι ανανεώσιμοι. πρώτη παρατήρηση λοιπόν ήταν αυτή. δεύτερη παρατήρηση. Φαίνεται να λέτε τουλάχιστον στην ε, εισήγησή σας ότι μπορεί να υπάρχει ένα είδος θεωρίας της ε, υποκατάστασης όταν ε, λείπει δηλαδή ένας, μια πρώτη ύλη. Παραδοσιακά αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να το εγκαταστήσουμε από μια άλλη πρώτη ύλη, μια άλλη τεχνολογία. Πιστεύετε ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε σε όλους τους τομείς. Τρίτη ερώτηση. Πιστεύω ότι για τις πρώτες ύλες και κυρίως για την ε, ιεραρχία της ε, εξάλληψης ή της μείωσης αυτών των πρώτων δεν είναι το ίδιο επίγον για όλες όσον αφορά την οικονομική χρήση και την αποτελεσματική τους χρήση. Το πετρέλαιο είναι η σπουδαιότερη πρώτη ύλη στον κόσμο και η εμπορική της αξία αντιστοιχεί στο σύνολο των υπόλοιπων πρώτων υλών παγκοσμίω. Και αυτό είναι που σιγά σιγά τελειώνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν όμως άλλες πρώτες ύλες που είναι λιγότερο σημαντικές από το πετρέλαιο. Και λέτε στην παράγραφο 19 ότι θα μπορούσαμε ίσως το 2020 να φτάσουμε σε ε, νέα χρήση 100% των πρώτων υλών. Πολύ καλό αυτό, αλλά αναφέρεστε και στο φόσφορο. Είστε βέβαιος ότι για το φόσφορο θα μπορούσαμε να φτάσουμε εύκολα το 100%? So the next speaker is Horst Schnellhardt afterwards Satu Ο Horst Schnellhardt και μετά η Satu Hassi. Ευχαριστώ πολύ. Έχει πολύ δύσκολο έργο ο εισηγητής. Έχουμε μείωση των πόρων στην Ευρώπη και στην ε, έκθεση αυτή δεν είναι ε, δυνατόν ε, να μπει κανείς σε λεπτομέρειες χωρίς να ξεχάσει τη συνολική εικόνα. Τα λέω λίγο προκλητικά. Υπερβάλλω λίγο τώρα στην αρχή, αλλά βλέπουμε ότι θα πρέπει οι επιδοτήσεις ε, ε, ότι οι περιβαλλοντικές ε, ενισχύσεις θα πρέπει μέχρι το 2020 να καταργηθούν. Θέλουμε μια γενική συζήτηση, αλλά μπαίνουμε αμέσως σε λεπτομέρειες η διαδικασία του ανταγωνισμού της συνεργασίας και της ανάπτυξης και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας την οποία ήδη έχουμε ε, ε, ξεφεύγει από τα πλαίσια. Ε, είναι λοιπόν πάρα πολύ δύσκολη η διαδικασία αυτή. Είτε θα παραμείνουμε γενικοί και δεν βρίσκω τόσο και στις πέντε προτεραιότητες, αν παραμείνουμε σε γενικό επίπεδο, αλλά υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα στην έκθεση όπου λέω ότι πρέπει να το σκεφτούμε, να σκεφτούμε σε τι βαθμό αυτό επηρεάζει τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων και πόσο επηρεάζει τη ζωή των πολιτών. Ε, να τους λέμε να τρώνε λιγότερη ζωική πρωτεΐνη. Ε, στην ε, Ανατολική Γερμανία επί κομμουνισμού υπήρχαν τέτοιες κατευθύνσεις, αλλά νομίζω πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην μπούμε σε τόσες λεπτομέρειες. ε, βρίσκω κάπως υπερβολικά ε, αυτά που αναφέρονται, ε, αλλά όσον αφορά το χρόνο. Δεν πρέπει να παραμείνουμε σε, ε, ε επίπεδο. Βρίσκω ότι είναι Πολύ σύντομες οι προθεσμίες και για την ε, υποβολή των τροπολογιών ε, και για την ε, ψηφοφορία. Δώστε μας περισσότερο χρόνο. Δεν, περιέχει πολύ σημαντικά θέματα η έκθεση αυτή. Δεν θα γίνουν λιγότερο σημαντικά αν βιαστούμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σνέλχαρτ. Δυστυχώς φάγαμε τη σειρά μια συναδέρφου και θα τη δώσουμε πρώτα το λόγο πριν το δώσουμε στη Σατουχάση. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ τον ε, εισηγητή για την πολύ καλά δομημένη έκθεσή του και για την ε, σαφή παρουσίαση. Εγώ βλέπω ως εξής την κατάσταση με τις πρώτες ύλες. Εάν κάποιος πάσχει από χρόνια ασθένεια, κάποιος που που θα αλλάξει την, ε, τον τρόπο ζωής του λόγω της χρόνια ασθένειάς του μπορεί να ζήσει περισσότερο από άλλου, αλλά θα πρέπει να αλλάξει τον τρόπο ζωής του, το τι τρώει κλπ. Το ίδιο ισχύει για τις πρώτες ύλες. Ε, αυτό πιο, πιο επώδυνο θα είναι να ε, έχουμε ανάπτυξη και να μειώσουμε την κατανάλωση των πόρων. Δεν υπάρχει πολύ κατανόηση από τους πολίτες Ευρώπης για το θέμα αυτό, ιδιαίτερα όχι όσον αφορά τον προσωπικό τρόπο ζωής τους. Και γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε στοιχεία στους ανθρώπους για να τους πείσουμε σε ατομικό επίπεδο. Και μιλάμε για μαζική πληροφοριακή εκστρατεία. Ε, πρέπει να καταναλώνουμε λιγότερο και να παράγουμε περισσότερο. Αυτά κατά κάποιο τρόπο ε, αντιφάσουν μεταξύ τους και όσον αφορά τα απόβλητα. Ε, εγώ βλέπω να υπάρχει σημαντική ευκαιρία τον οικολογικό σχεδιασμό. Ο οικολογικός σχεδιασμός μπορεί να αποτελεί σημαντική πηγή καινοτομίας και εάν δεν σχεδιάζονται έτσι τα προϊόντα ώστε δηλαδή να είναι κατά 100% ανακυκλώσιμα, θα υπάρχει σύγχυση όσον αφορά ε, τα απόβλητα. Το θέμα της τιμής είναι επίσης επώδυνο. Όπως άλλωστε είναι επώδυνο και το θέμα της φορολογίας. Ε, συμφωνώ με τους συναδέλφους μας ότι κατά την ε, κρίση αυτή... Τρει σύντομε παρατηρήσει. Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για, ένα, για το πολύ καλό του σχέδιο έκθεσης. Έπειτα, πρώτη παρατήρηση. Έμαθα κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομία μου στην πολιτική ότι πολύ συχνά ότι ό,τι δεν συνοδεύεται από δεσμευτικούς στόχους δεν ε, μένει μόνο στα λόγια. Οπότε οι στόχοι και οι δείκτες ε, είναι, οι δεσμευτικοί στόχοι και οι δείκτες είναι πολύ σημαντικό, ε, προς σημαντική προτεραιότητα. Έπειτα, πρέπει να με φροντίσουμε ώστε οι πολιτικές της Ένωσης και κυρίως οι καινούργιες πολιτικές να μην μας φέρουν, να μην μας οδηγήσουν σε άλλη κατεύθυνση από την βελτίωση της χρήσης των πόρων. Ήδη έχω αναφέρει την βιομάζα και εκεί θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε οι πρόσφατες μας πολιτικές να μην επιδεινώσουν την αποδοτικότητα των πόρων. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα για το γεγονός ότι το, για, την, για την χρήση των πόρων εκεί όπου έχουμε την καλύτερη απόδοση του συγκεκριμένου υλικού. Αυτή θα πρέπει να είναι μια αρχή που μας, θα μας καθοδηγεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, κατασκευή σπιτιών, κατασκευή επίπλων από το ξύλο, και όχι καύση του ξύλου. Δεν έχω χρόνο για το τρίτο σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο Ρίχαρτ Ζήπερ και κατόπιν ο άτομ Κέρεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή για την έκθεση που έχει υποβάλει. Ωστόσο θα ήθελα να θυμίσω ότι δεν με, ζούμε σε ένα νησί στην Ευρώπη. Υπάρχει ο διεθνής ανταγωνισμός. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ε, τι ε, μηνύματα ε, στέλνουμε στον τομέα της φορολογίας, για παράδειγμα. Η ανθρώπινη εργασία είναι ο παράγοντας που πιο δύσκολα που μπορεί να μεταφερθεί ε, αεροπορικά. Ε, θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να ε, αποφύγουμε την, αποτρέψουμε την μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων εκτός Ευρώπης και να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τους χώρους παραγωγής στην Ευρώπη και να πετύχουμε τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα. Η έκθεση... Η έκθεση αυτή μου θυμίζει αυτό που είπε ο Διευθυντή του Γραφείου Ευρυστεχνιών της ε, Αμερικής το 1869, ότι όλες οι βασικές ε, εφευρέσει ήδη έχουν γίνει. Ε, ο συνάδελφος από την από τους πράσινους ε, αναφέρθηκε στο θέμα ε, ανανεώσιμος μη ανανεώσιμος. Ε, ας κοιτάξουμε για παράδειγμα την ικανότητα των υπολογιστών μας. Σκεφτείτε την, την αύξηση που βλέπουμε θα πρέπει να αποφύγουμε να πετύχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Όσο καλύτερα καταλάβουμε τους πόρους μας, όσο καλύτερα τους ε, ε, διακρίνουμε και τους καταλήμουμε, τόσο ε, καλύτερα θα είναι. Και είναι πολύ σημαντική η διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Άνταμ Κέρεκ. Σας ευχαριστώ. Από τις πέντε προαναφερθήσεις ε, προτεραιότητες, περισσότερο μου αρέσει η δεύτερη προτεραιότητα ε, για την αγορά των δευτερογενών ε, υλών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δυστυχώς μηχανισμούς της αγοράς που να ενεργοποιήσουν την αξιοποίηση αυτών των υλών. Δυστυχώς δεν υπάρχουν κίνητρα, οικονομικά κίνητρα για την ε, διεξαγωγή καινοτόμων ερευνών για την αξιοποίηση αυτών των ε, υλών, των πρώτων υλών. Θα μπορούσαμε λοιπόν ε, να υποβάλουμε και προτάσεις. Τι μηχανισμούς στην αγορά ξέρουμε. Δυστυχώς οι φθηνές πρωτεσίλες είναι παρελθόν. Οι Κινέζοι μας έδειξαν ότι ε, δεν πρόκειται να μας πουλήσουν πολλές σπάνιες ε, γέες ή σπάνιες πρώτες ύλες. Οι Ρώσοι προς το παρόν μας πουλάνε, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι στο μέλλον ε, δεν θα έχουμε πρόβλημα ανεφοδιασμού και εξαιτίας της σπάνιας, της έλλειψης. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσει η Ευρώπη να εξασφαλίσει δικές της πρώτες ύλες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτή είναι πολύ σημαντική προτεραιότητα. Να μπορέσει η Ευρώπη να αξιοποιήσει τις δικές της πρώτες ύλες, τις δικούς της πόρους και φυσικά μια ισορροπημένη οικονομία, ε, μια οικονομία που θα αξιοποιεί αρθολογικά στους πόρους, δεν είναι μια άπλιστη και πλέον εκτική οικονομία. Μερικές φορές μπορούμε με τοπικές πρωτεσίλες ε, να καλύψουμε τις ε, κατασκευαστικές μας ανάγκες, τις ανάγκες κατασκευής αυτοκινητοδρόμων σε τοπικό επίπεδο αλλά θα πρέπει να κινητοποιήσουμε τον τοπικό πληθυσμό για τα θέματα αυτά, για την αξιοποίηση αυτών των πόρων. Γιατί οι τοπικές κοινότητες ε, ε, αναλαμβάνει και το περιβαλλοντικό κόστος και το κοινωνικό κόστος ε, και το οικολογικό. Γιατί λοιπόν να μην προσθέσουμε και αυτό το σημείο της κινητοποίησης των τοπικών πληθυσμών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στην Κομισιόν. Στην Κάριν Φόβελ, παρακαλώ. Um, Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό το σχέδιο έκθεσης. Βρίσκουμε ότι υποστηρίζει πολύ και αντικατοπτρίζει το δική μας σκέψη και το επίπεδο φιλοδοξίας στο θέμα της καλύτερης χρήσης των πόρων. Πολλές προτάσεις γίνονται στην έκθεση αυτή, σίγουρα θα τις εξετάσουμε. και φυσικά θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με βάση τους πόρους και τις δομές που έχουμε τώρα και βέβαια να δούμε πού θα μπορούσαμε να έχουμε ακόμη περισσότερες φιλοδοξίες. Πολλή δουλειά ήδη γίνεται σε αυτόν τον τομέα, ε, όπως το Ευρωπαϊκό Εξάμενο, όπου έχει ενταχθεί το θέμα της καλύτερης χρήσης των πόρων όπως ε, περιβαλλοντικές, μέσω περιβαλλοντικών επιδοτήσεων αλλά και μέσω της ε, της δυναμικής ανάπτυξης της ανακύκλωσης, για παράδειγμα. Θεωρούμε πως είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλα αυτά τα θέματα, αλλά σίγουρα θα υπάρξει κάποιο παζάρεμα σε σχέση με την ταχύτητα και την ε, εμπλοκή των ενδιαφερομένων φορέων. Υπάρχει επίσης στήριξη για τη βιώσιμη κατανάλωση της παραγωγής. Σκοπεύουμε να κάνουμε μια ανακοίνωση για το πρασίνισμα της ενιαίας αγοράς μέχρι το τέλος του έτους. Θα είναι ένα από τα εργαλεία, από τα μέσα εφαρμογής ε, της ε, αποτελεσματική χρήση των πόρων στον το τομέα και εκεί θα συμπεριλαμβάνονται διάφορες δράσεις για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για το πρασίνισμα της νέα αγορά και θα αναφέρονται και κάποια θέματα που αναφέρονται και σε αυτή την έκθεση όπω οι κρατικέ προμήθειε, ε, το, αποτύπωμα, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα κτλ. Η πίνακα επιδόσεων και γίνεται αυτή τη στιγμή δημόσια διαβούλευση μέχρι τι 3 Απριλίου. Θεωρούμε πω είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη συλλογή απόψεων και επιπλέον πληροφοριών που τροφοδοτούμε αυτήν την διαδικασία με όλες αυτές τις πληροφορίες ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ευρύτερες ανάγκες του κοινού. Σε σχέση με τους στόχους θα χρειαστούν πολύ έντονες προσπάθειες από τα κρατημέλη. Θα τα αναλύσουμε όλα αυτά εις βάθος το 2013 όταν θα εξεταστούν οι στόχοι των οδηγιών για τις χωματερές και τη διαχείριση των αποβλήτων ε, όσον αφορά την ιδέα για τη δημιουργία ενός χώρου Σέγγεν για τα απόβλητα ε, προσπαθούμε να συμβάλλουμε σε αυτό το στόχο αναπτύσσοντας κριτήρια ε, για τα απόβλητα που θα ίσιαν για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας περί αποβλήτων σε ολόκληρη την Ένωση παίζει ρόλο κλειδί εδώ. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την υποστήριξή σας. Προσβλέπουμε στην συνέχιση της στενής μας συνεργασίας ε, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με την εφαρμογή του οδικού χάρτη. Ευχαριστώ την Κομισιόν. Ε, τελευταίος έχει το λόγο ο μιλητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, για την ευρεία υποστήριξή τους ω προς το γενικό μήνυμα της έκθεσης αυτής. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Δεν ε, θα πω σε λεπτομέρειες ε, για τα πολλά θέματα που τέθηκαν. Ε, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι πολλά από τα θέματα που θίξατε ήδη τα έχω στο ράφι με τις τροπολογίες μου. Χρειάζομαι όμως τη βοήθειά σας για να γίνει πιο φιλόδοξη και πιο ισχυρή η έκθεση αυτή. Προσβλέπω λοιπόν ε, στις ε, ε, συνεισφορές σας. Κάποια στοιχεία που έθιξαν αρκετοί από εσά. Καταρχήν, έχουμε την ιδέα ενός χώρου Σέγγεν για τα απόβλητα. Το έχω συζητήσει αυτό με πολλούς. Σκέφτηκα να αλλάξω όνομα, να μιλάω για εσωτερική αγορά ε, αποβλήτων. Μ' αρέσει όμως ε, η ιδέα του Σέγγεν, διότι η ιδέα είναι τα κράτη-μέλη που είναι έτοιμα να μπορούν να συμμετάσχουν και το ίδιο ισχύει και για τα απόβλητα. Συμφωνώ απόλυτα με κάποιους από τους συναδέρφους που έθιξαν το θέμα αυτό. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ανάπτυξη Τη ε, πολιτική αποβλήτων τους. Ε, κάποια κράτη-μέλη δεν είναι έτοιμα ακόμα να συμμετάσχουν ε, σε έναν τέτοιο χώρο. Και δεν είμαι υπέρ του να μεταφέρουμε τα απόβλητα όσο περισσότερο μπορούμε στην Ευρώπη. Του αντίον πιστεύω ότι θα πρέπει να διαχειριζόμαστε τα απόβλητα εκεί όπου παράγονται. Εάν Ε, είναι δυνατόν ε, να γίνει η διαχείρισή τους σε κάποια βασικά σημεία της Αυτό θα είναι καλό και γι' αυτό ε, υπέβαλα αυτή την ιδέα για μια περιοχή Σέγγεν. Βλέπουμε επαναστατικέ εξελίξεις στον τομέα των αποβλήτων. Αν δείτε τα επενδυτικά κεφάλαια που επενδύονται στην διαχείριση αποβλήτων, βλέπουμε ότι μετατρέπεται ο τομέας από μια εντό εισαγωγικών βρώμικη δουλειά σε, μια, σε έναν πολύ επαγγελματικό και κερδοφόρο τομέα. Ε, και όπως πολύ σωστά υπόθηκε, δεν, δεν είναι απαραίτητα απόβλητα, είναι πολύτιμος πόρος. Η τιμολόγηση είναι άλλο θέμα. Φοβάμαι ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να ε, διαφωνούμε όσον αφορά τον καλύτερο τρόπο. Εγώ εδώ προτιμώ να μην εισάγω έναν ε, φόρο ε, πρώτων υλών. Διότι κοιτάξτε πόσο αυξάνονται οι τιμές των πρώτων υλών. Ε, δεν χρειάζεται φορολογία για να ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις να αρχίσουν να ανακυκλώνουν τα υλικά τους. Τα δευτερεύοντα υλικά θέλουμε να τα προωθήσουμε για τους λόγους που σας ανέφερα πριν. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να ε, κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα σε διάφορους ε, πόρους. Οι ιδιωτικοί πόροι είναι σημαντικό πρόβλημα, είναι υπερβολικά ε, φτηνοί και η χρήση Ε, η ζημιά που κάνουν ε, στον ε, στο περιβάλλον και στη βιοπικιλότητα δεν αντικατοπτρίζεται στην τιμή. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε πέρα από το ΑΕΠ και ο τρόπος υπολογισμού τους σίγουρα θα αποτελέσει βήμα προόδου. Κάποιος είπε ότι δεν ζούμε στην, σε ένα νησί στην Ευρώπη, θα πρέπει να κοιτάξουμε τον ανταγωνισμό μας με τον υπόλοιπο κόσμο. Συμφωνώ απόλυτα. Και γι' αυτό προτείνω αυτά που προτείνω. Γι' αυτό ακριβώς όταν συνέταξα την ε, έκθεση, σκέφτηκα γιατί είναι η ΕΝΒΗ επί της ουσίας αρμόδια και όχι αυτή των οικονομικών θεμάτων. Εάν κοιτάξετε την αύξηση των τιμών για τις επιχειρήσεις, για τις πρώτες ύλες, θα δείτε ότι η αύξηση είναι τεράστια. Είναι τώρα ε, η εποχή των ε, ετησίων ισολογισμών των εταιριών και αν κοιτάξετε τις τιμές των πρώτων υλών θα δείτε ότι αγωνίζονται οι επιχειρήσεις ε, να καλύψουν το κόστος. Ε. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι, κοινός, ότι δημόσιος και ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να συνεργαστούμε ώστε η Ευρώπη να ε, γίνει η περιφέρεια του κόσμου που διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά τους πόρους και έτσι να γίνει και η πιο ανταγωνιστική σε έναν από τους πιο βασικούς τομείς της πολιτικής ανταγωνισμού αυτή τη στιγμή όχι μόνο δηλαδή απλά γνωρίζω απόλυτα το θέμα του, ανταγωνιστού, πιστεύω, του ανταγωνισμού, πιστεύω ότι είναι ζωτική σημασία στην όλη συζήτηση και θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό. Όσον αφορά την ανθρώπινη διατροφή. Εγώ είμαι από την ομάδα των φιλελευθέρων και το έχω συζητήσει αυτό στην ομάδα μου. Το τι θα τρώει ο καθένα, θα το αποφασίζει ο καθένα αν θέλει να τρώει κρέα ή όχι. Και συμφωνώ με αυτό από την άλλη, δεν θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο να μην μπορούμε να συζητήσουμε ως πολιτικοί. Γνωρίζουμε ότι τις επόμενες ε, δεκαετίες θα πρέπει να τρώμε λιγότερο κρέας ανά άτομο. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο το γνωρίζουμε σίγουρα. Γιατί λοιπόν να μην ε, αρχίσουμε ε, ήδη μια συζήτηση και όχι να αναγκάσουμε τον κόσμο να αλλάξει τη διατροφή του, αλλά να γνωρίζει καλύτερα τι, τι τρώει και για λόγους υγείας. Πρόεδρε, η κυρία Μέξης μόλις έφυγε, θα συζητήσω λοιπόν μερό το θέμα μαζί της. Νομίζω ότι κάλυψα τα περισσότερα από τα θέματα που θύχτηκαν. Αναφέρθηκε η διάκριση ανάμεσα στις ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες ε, πρώτες ύλες. Ε, μου αναφέρατε το νερό ως παράδειγμα. Ε, είναι όμως πρόβλημα το νερό, παρότι είναι ανανεώσιμο, ανανεώσιμος πόρος. Και όταν ε, μιλάμε για την καλύτερη αποτελεσματικότητα των πόρων, δεν μπορούμε να έχουμε μια λύση που να ισχύει για όλα. Ε, και ακόμα και οι διαφορές μεταξύ περιφερειών, και ακόμα και εντός του ιδίου κράτους μέλους, είναι μεγάλες και θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας αυτά. Ξέρουμε ότι σε κάποια κράτη-μέλη καλύτερο να χρησιμοποιεί κανείς ε, λιγότερο νερό. Πολλά από αυτά τα κράτη-μέλη ήδη έχουν σχετικές πολιτικές όπως η Ισπανία. Άλλα κράτη-μέλη όπως το δικό μου, οι κάτω χώρες έχουν αρκετό νερό. Ε, έχουμε πρόβλημα όμως με την ποιότητα του νερού. Μερικές φορές λοιπόν το πρόβλημα είναι η ποιότητα, άλλες φορές είναι η ποσότητα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα δύο. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι κάλυψα αρκετά από τα θέματα που ανέφεραν οι συνάδελφοι. Ε, προσλέπω στις ε, προτάσεις σας ε, για να βελτιώσουμε την έκθεση και σας ευχαριστώ για την ευρία υποστήριξή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε Γκερμπράντη. Ε, που απαντήσατε στα, στις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις. Είναι σημαντική η έκθεση αυτή. Φυσικά ο καθένας θέλει να δει να αντικατοπτρίζονται οι ιδέες του σε αυτήν, ε, αλλά Είδαμε ότι ήδη με τις ε, πέντε προτεραιότητες ε, θα είναι δύσκολο να βρούμε συμφωνία. Σας παρακαλώ λοιπόν ε, κατά την ψηφοφορία να είσαστε συγκεντρωμένοι ώστε να καταλήξουμε στο σωστό αποτέλεσμα όσον αφορά τις προθεσμίες και το χρονοδιάγραμμα σε συμφωνία με τον εισηγητή έχουμε θέσει την προθεσμία για τις τροπολογίες στις 8 Μαρτίου. Παρατείναμε δηλαδή την προθεσμία. Στην Επιτροπή ΕΝΒΗ θα ψηφίσουμε στις 26 Απριλίου και στην Ολομέλεια του Μαΐου θα ψηφίσουμε οριστικά το, την έκθεση αυτή. Ε, κύριε Σνέλχαρτ, να σας καθησυχάσω. Έχουμε παρατείνει τη διαδικασία την προθεσμία συγγνώμη, για τις τροπολογίες. Ωραία, έτσι ολοκληρώσαμε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Πρόκειται για έκθεση εμπειρογνωμόνων ε, ενσωμάτωση της αεροπορίας στο σύστημα εμπορίας εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ήδη έχουν ζητήσει αρκετοί το λόγο. Έχει περάσει αρκετός χρόνος από τότε που λάβαμε σχετική απόφαση. Αλλά ε, για την εφαρμογή των ε, θεμάτων αυτών ε, δεν είμαστε μόνοι μας και γι' αυτό θέλω μια έκθεση εμπειρογνωμοσύνης από την Κομισιόν σχετικά με το πόσο έχει προχωρήσει η νομοθεσία αυτή. Ακούμε ειδήσει σε άλλα μέρη του κόσμου Αναφέρεται το θέμα των ευρωπαϊκών αεροπλάνων. Ε, περιμένω λοιπόν με αγωνία να ακούσω τι έχει να μας πει η Κομισιόν. Παρακαλώ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θερμές ευχαριστίες για την ε, δυνατότητα που μας δίνετε και την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε για τις τελευταίε εξελίξει ό,τι αφορά τη συμπερίληψη της αεροπορία στο σύστημα εμπορίας εκπομπών. Δυστυχώ, η συμπερίληψη της αεροπορία στο σύστημα εμπορίας εκπομπών προσκρούει διεθνώ σε πολύ σημαντικέ αντιστάσεις. Πολύ συχνά αναφέρεται στη διασκέψη κορυφής τρίτων χωρών, πρόσφατα στη Μόσχα για παράδειγμα, εξετάστηκε. Αλλά σίγουρα πιστεύουμε κύριε Πρόεδρε ότι η καλύτερη λύση είναι ο διάλογος σε διμερές και πολυμερές επίπεδο. Η Ευρώπη ήταν ανέκαθεν αναφανδόν υπέρ ε, παγκοσμίων δράσεων, σφαιρικών δράσεων για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών που ούτως ή άλλως τις βιώνουμε παγκοσμίως. Εμείς ήδη αποφασίσαμε να ενσωματώσουμε την αεροπορία στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Υπομόνων και θεωρούμε ότι ή άλλως τις βιώνουμε παγκοσμίω. Εμείς ήδη αποφασίσαμε ε, να ενσωματώσουμε την αεροπορία στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών και θεωρούμε ότι το, ε, η Διεθνής, αεροπορία, η Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας, η ΚΑΟ των Ηνωμένων Εθνών, τάχθηκε υπέρ αυτής της πολιτικής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που ανάγεται ήδη στο 2004. Από τότε λοιπόν η ΚΑΟ αποφάσισε να μην θεσπίσει ένα νέο παγκόσμιο σύστημα εκπομπών αερίων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, αλλά να επικεντρωθεί σε άλλα μέτρα, όπως εφαρμογή μέσω της συμπερίληψης ε, σε κρατικά ή περιφερειακά συστήματα εμπορίας εκπομπών. Θεωρούμε όμως ότι οι δράσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εσωμάτωση αεροπορία στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου συνάδει πλήρως με την ε, προσέγγιση της ΙΚΑΟ από το 2004. Τώρα, άσχετα με το ιστορικό αυτό, αν κάποια χώρα του κόσμου ή κάποιες χώρες του κόσμου είναι έτοιμες ε, και ε, στενιστούν μια φιλόδοξη παγκόσμια προσέγγιση της ΕΚΑΟ, έστω και τώρα, εμείς είμαστε οι πρώτοι που θα επικροτήσουμε μια τέτοια συμπεριφορά. Η δράση όμως θα πρέπει να προωθεί μέσω της ΕΚΑΟ, ε, με μέτρα που θα στηρίζονται στην αγορά για να μειωθούν οι εμπορίες εκπομπών της διεθνούς πολιτικής αεροπορίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα αφιστεί προσπαθειών και θα επιδιώξει κάποιε πρωτοβουλίε και θετικά βήματα για να ενταχθεί το θέμα τη εμπορία εκπομπών τη πολιτική αεροπορία της αεροπορίας στο πλαίσιο τη ΙΚΑΟ. Από αυτή την άποψη, στην διάσκεψη κορυφή με τι ΗΠΑ το περασμένο Νοέμβριο, είχαμε την ευκαιρία να διατρανώσουμε την κοινή μα δέσμευση για σημείωση πρόοδου σε αυτό τον οργανισμό του ΙΕ για την ε, πολιτική αεροπορία των ΕΚΑΟ. Πρόσφατα, ο πρόεδρος του ΕΚΑΟ, κ. Γκόμπε, εγκινήσε μια πρωτοβουλία καλώντας τις χώρες να εξετάσουν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις και μέτρα που θα στηρίζονται στην αγορά στο πλαίσιο της ΕΚΑΟ. Εμείς είμαστε υπέρ φυσικά μιας τέτοιας προσέγγισης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει ενεργά στην πρωτοβουλία της ΕΚΑΟ και μάλιστα έχει συστηθεί και μια ομάδα εργασίας ε, σε αυτό τον οργανισμό του ΟΗΕ, τον ΙΚΑΟ, προκειμένου να εξεταστούν ε, μέτρα που θα στηρίζονται στην αγορά. Ο ΙΚΑΟ θα υποβάλει προτάσεις μέχρι τα τέλη του έτους και είναι πολύ σημαντικό και για τη σημερινή μας συζήτηση εδώ. Τώρα, για παγκόσμια δράση με μέτρα που θα στηρίζονται στην αγορά, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε τρία πολύ σημαντικά στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι οτιδήποτε συμφωνηθεί για μέτρα που θα στηρίζονται στην αγορά στην ΕΚΑΟ θα πρέπει να οδηγηθούν σε μείωση των εκπομπών σε σχέση με τα υφιστάμενα μέτρα. Ακόμη και από τις 30 χώρες που εφαρμόζουν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών. Δεύτερον, το σύστημα της ή που εφαρμο... το σύστημα που θα εφαρμοστεί από τις χώρες δεν θα πρέπει να ε, θεσπίζει διακριτική μεταχείριση βάρος κάποιων αεροπορικών εταιριών γιατί η αποφυγή της διακριτικής μεταχείρισης είναι βασική αρχή της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού για τις, αεροπορία, για τις αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε μια ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά. Τρίτο στοιχείο, ένα στεναρό παγκόσμιο σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει, να περιλαμβάνει στόχους και μέτρα για τα μέλη της ΕΚΑΟ. Και για να είναι ένα παγκόσμιο σύστημα αποτελεσματικό και όντως να συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών, θα πρέπει να στηρίζεται σε μια συμφωνία για τους στόχους και για αποτελεσματικούς τρόπους ε, υλοποίησης αυτών των στόχων. Πολλές χώρες προετοιμάζουν ε, σχέδια δράσης που θα υποβάλουν ε, στη Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας μέχρι τον Ιούνιο και έτσι οι χώρες ε, θα συμβάλλουν στην πρόταση αυτή. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά σε ό,τι αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις για την Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών λειτουργεί πια εδώ και 8 χρόνια. Οι αερογραμμέ ε, προσχώρησαν πλήρω στο σύστημα αυτό τον Ιανουάριο και έχουμε μάθει πολλά από αυτή την εμπειρία, την πολιτή μα εμπειρία και πολύ ευχαριστώ θα μοιραστούμε τα πορίσματα αυτή τη εμπειρία ε, στην διαδικασία που ξεκίνησε στην ΙΚΑΟ. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για το Σύστημα Εμπορία Εκπομπών που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο το 2008 ε, έχει μεγάλη σημασία για μας. Η νομοθεσία αυτή στηρίχθηκε σε, μία, σε αποφάσεις ε, που συνέχισαν ε, την Γενική Συνέλευση της ΙΚΑΟ του 2004 και όπως είπα φυγραμμίζονται πλήρως με την προσέγγιση που εφάρμοσε τότε, που υιοθέτησε τότε η ΙΚΑΟ. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών και Σχετική Νομοθεσία περιλαμβάνει πολύ σημαντικές διατάξεις περιελαστικότητας και θα ήθελα εδώ να σταθώ σε αυτές τις δύο πολύ σημαντικές διατάξεις περιελαστικότητας. Καταρχήν, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει τη δυνατότητα αποκλεισμού ε, ε, πτήσεων που έρχονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, με βάση τη δράση των τρίτων χωρών για να περιορίσουν τι κλιματικές αλλαγές που οφείλονται στην αεροπορία. Φυσικά αυτό γίνεται χωρίς διάκριση και ισχύει και για τις ε, πτήσεις ευρωπαϊκών και για τις πτήσεις μη ευρωπαϊκών εταιριών που έρχονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερο σημαντικό μέτρο ελαστικότητα που περιλαμβάνεται στην κοινοτική νομοθεσία προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλήρω αφοσιωμένη και δεσμευμένη να συνεχίσει τις προσπάθειές της για να σημειωθεί πρόοδος διεθνώς ε, στην ΙΚΑΟ για να περιοριστεί ο κλιματικός αντίκτυπος της αεροπορίας και να μπορέσουν οι αερογραμμές ε, να αναπτυχθούν με βιώσιμο τρόπο. Σε περίπτωση σύναψης παγκόσμιας συμφωνίας για διεθνή μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της αεροπορίας, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει αναθεώρηση ε, και τροποποίηση αντίστοιχα του συστήματό τη. Φυσικά σε μια ενδεχόμενη τέτοια διαδικασία το Κοινοβούλιο θα ανανοιχθεί όπω προβλέπεται. Θα ήθελα στη συνέχεια να σα κάνω μια ενημέρωση για τι ε, διμερεί μα συζητήσει και τι πολυμερεί συζητήσει που γίνονται για το θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγης ε, την κατάσταση και των χωρών που έχουν δηλώσει επιφυλάξει αλλά και των χωρών που ενδιαφέρονται για διάλογο. Όπως θα ξέρετε, στη διάσκεψη κορυφής με την Ινδία και την Κίνα πρόσφατα αλλά και πέρυσι με τις Ηνωμένε Πολιτείε και τη Ρωσική Ομοσπονδία το σύστημα της ε, αεροπορίας ήταν στην σε διάταξη. Πιστεύουμε ότι ο σωστός τρόπος για να υπερκεραστούν οι διαφωνίες και οι διαφορές είναι ένας επικοδομητικός και καρποφόρος διάλογος σε διμερές αλλά και πολυμερές επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες των διεθνών μας εταίρων και ενθαρρύνουμε έναν εργοδιάλογο με κυβερνήσεις τρίτων χωρών προκειμένου να δούμε τι πρόοδο σημειώνεται στην ΕΚΑΟ και ε, υπό το φως των ε, διατάξεων περί ελαστικότητας της κοινοτικής νομοθεσίας. Σε ό,τι αφορά την ε, διάσκεψη κορυφής της Μόσχας που έλαβε χώρα 21 και 22 Φεβρουαρίου. Εκεί ε, συμμετείχαν πολλές χώρες και θέμα της συζήτησης ήταν η συμπερίληψη της αεροπορίας στο σύστημα εμπορίας εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η δήλωση που απέρευσε από τη διάσκεψη αυτή κορυφής ήταν πολύ ευπρόσδεκτη, γιατί περιλαμβάνει το ενδιαφέρον των χωρών αυτών για περαιτέρω επεξεργασία των προτάσεων της ΙΚΑΟ και νομίζω ότι αυτό το μήνυμα ήταν πολύ σημαντικό, το μήνυμα της διάσκεψης κορυφής της Μόσχας. Χαιρόμαστε επίσης γιατί ε, οι χώρες που συμμετείχαν στη διάσκεψη της Μόσχας αναγνώρισαν ότι ο περιορισμός ε, εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου είναι προτεραιότητα. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η βούληση που εκδηλώθηκε να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες θετικέ και επικοδομητικές προτάσεις ε, που θα, προταθούν, θα υποβληθούν στην ΙΚΑΟ προκειμένου να διαθετήθει παγκόσμια δράση κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως σας είπα. Είναι και η ώρα να αναλάβουν όλες οι χώρες σοβαρές δεσμεύσεις για μια φιλόδοξη παγκόσμια συμφωνία και επίσης να είμαστε πολύ ακριβείς και συγκεκριμένοι για τους στόχους μας και πότε θα τους υλοποιήσουμε. Ανάλογα με το κατά πόσο θα... μέχρι μάλλον μέχρι ότου εφαρμοστεί αυτή η παγκόσμια η συμφωνία, το ευρωπαϊκό σύστημα για την συμπερίληψη αεροπορίας θα ισχύει για όλες τις ε, αεροπορικές εταιρείες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πέρυσι το Δεκέμβριο ενέκρινε αυτή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπα όμως ήδη, και νομίζω ότι ήμουν σαφέστατη, η νομοθεσία αυτή, η κοινοτική νομοθεσία προβλέπει δύο σημαντικά μέτρα ελαστικότητας που δεν είναι εξαντλητικά. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που μας δίνει η νομοθεσία για να προωθήσουμε την σύναψη και παγκόσμια συμφωνίας. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι υπάρχει ανάγκη για ένα προβλέψιμο μακροπρόθεσμο παγκόσμιο πλαίσιο για να περιορίσουμε τις εκπομπές αεροθερμοκηπίου από την αεροπορία και γι' αυτό χρειαζόμαστε μέτρα που θα στηρίζονται στην αγορά. Είναι απαραίτητο στοιχείο μιας συνολικής πολιτικής. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών είναι καταλήτης ε, για την παγκόσμια δράση και δεν ε, γύρει εμπόδια για μια τέτοια παγκόσμια δράση σε καμία περίπτωση. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών περιλαμβάνει και κάποιε ρήτρε ελαστικότητας που μπορούμε να τι αξιοποιήσουμε και διεθνώ αλλά και, και συγγνώμη, και πολυμερό. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τι διμερεί διαπραγματεύσει με όλε τι ενδιαφερόμενες χώρε, αλλά παρόλα αυτά πιστεύουμε ότι η διεθνή Οργάνωση πολιτική Αεροπορία είναι το κατάλληλο πλαίσιο για την ανέβρεση μια παγκόσμια λύση. Είμαστε υπέρ τη διαδικασία τη ΙΚΑΟ, που εγκαινιάστηκε πρόσφατα, όπω σα είπα, από τον πρόεδρο τη οργάνωση αυτή και επιθυμούμε την επιτάχυση της ε, δράσης προκειμένου να υιοθετηθούν κάποια μέτρα που θα στηρίζονται στην αγορά. Θα συνεχίσουμε την ενεργό συμμετοχή μας και τη συνεργασία μας με όλες τις χώρες που ενδιαφέρονται για την ανέβρεση μιας παγκόσμιας λύσης. Βέβαια, μια ε, παγκόσμια δράση που δεν θα, είναι, δεν θα δημιουργεί διακρίσεις θα είναι επωφελής για όλους μας, πιστεύω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την εισήγηση και επίσης διότι μας ξεκαθαρίσατε πού βρίσκεται η κατάσταση όσον αφορά το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Τώρα θα πρέπει να πω ότι έχουμε πολλούς ομιλητές και φυσικά όλοι θέλουν να πάρουν το λόγο. Οπότε παρακαλώ να τηρήσετε το όριο του 1,5 λεπτού. Ξέρω πως είναι πολύ φιλόδοξο. Δίνω το λόγο στους εισηγητές, μετά στον εισηγητή, μετά στους σκιώδη εισηγητή και μετά στους άλλους ομιλητές. Ο Πίτερ Λίζε. Σας ευχαριστώ πολύ. Την Επιτροπή και τον Πρόεδρο. Θα ήθελα να στηρίξω την Επιτροπή γιατί πρέπει να εφαρμόσουμε αυτή την νομοθεσία και όταν μιλάμε για ε, ευελιξία θα πρέπει να είναι αυτή η οποία προβλέπεται εντός της νομοθεσίας. Αν θέλουμε όντως να πετύχουμε κάτι με τρίτες ε, χώρες θα πρέπει να έχουμε <coughs> εξαιρέσεις για τις εισερχόμενες πτήσεις αλλά που να μην ε, δημιουργούν διακρίσεις. Θα πρέπει να ζητήσουμε από την Κομισιόν να επιβεβαιώσει ότι ορισμένοι μύθοι θα πρέπει να αναιρεθούν. Μιλάμε για τεράστιο φόρτο, γιατί έχει υπολογιστεί πως ε, για κάποια πτήση θα πρέπει να πληρώσει κανείς ακόμα 25 cents για το ETS και εθνική φορολογία μετά και δεν μιλάμε πραγματικά για τεράστιο φόρτο, μιλάμε απλά για τεράστια συζήτηση. Δώσε, δώστε μας νούμερα. Αυτό θέλω να ζητήσω από την Επιτροπή. Γιατί έχει γίνει αυτό το πολιτικό, δημιουργηθεί αυτό το πολιτικό θέμα, επειδή η Ένωση θέλει να δράσει εντός και εκτός Ένωσης ο κόσμος πιστεύει ότι δεν θα πρέπει να θεωρούμε τόσο σοβαρή την νομοθεσία μας όσο στη ΣΥΠΑ ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Και έπειτα το θέμα του κατά πόσο παίρνουμε στα σοβαρά τα κλιματικά θέματα ή όχι. Εγώ έχω συζητήσει με Αμερικανούς συναδέλφους και μιλούν για απαγορεύσεις, θέλουν να απαγορεύσουν τις αμαρικές, θέλουν να απαγορεύσουν τη συμμετοχή των αμερικανικών εταιριών σε αυτό το ETS. Ε, δεν πέρασε ποτέ αντίστοιχο σύστημα στη Γερουσία, από τη Γερουσία. Αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει η Κομισιόν και ότι αυτή η απαγόρευση δεν πέρασε στην ε, Γερουσία. Ευχαριστώ, κύριε Λίζε. Και τώρα με μεγάλη μου χαρά θα δώσω το λόγο στον Ματίας Χρότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ήμουν σκιώδης εισηγητής για το θέμα αυτό. Είχαμε μια συντριπτική πλειοψηφία εδώ στο Κοινοβούλιο που ψήφισε υπέρ αυτής της νομοθεσίας. Υιοθετήθηκε ομόφωνα στο Συμβούλιο και ε, σήμανε μια σημαντική ε, συμβολή. Ε, είναι ένα πραγματικό μέτρο θα βαθμολογηθούμε για το κατά πόσο μπορούμε να επιμείνουμε για την συμπερίληψη της αεροπλοείας στο ETS. Θα αφήσουμε να μας παρασύρει ο άνεμος. Όχι. Εγώ πιστεύω θα πρέπει να αντισταθούμε. Η διεθνής αεροπλοεία είναι διεθνής business. Η ΚΑΟ είχε 20 χρόνια τη συζήτηση αυτή και δεν προέβη ποτέ σε δράση. Η Ευρώπη αποφάσισε να ενεργήσει ως νομοθέτης, λάβαμε απόφαση και οφείλουμε να ασκήσουμε πιέσεις ώστε να αναλυφθούν δράσεις σε διεθνές επίπεδο, στην ΕΚΑΟ. Κάναμε εκεί αυτό που έπρεπε θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οποτεδήποτε μια κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία συνομιλεί με άλλε κοινοβουλευτικέ αντιπροσωπείες σε ολόκληρο τον κόσμο θα μιλά και για αυτό εδώ το θέμα. Θα έχει αυτό το θέμα στην ημερήσια της διάταξη. Καλύτερο τρόπο θα ήταν η φορολόγηση, θα χρειαζόταν ομοφωνία για την εμπορία εκπομπών ήταν η καλύτερη λύση, δεν δημιουργεί διακρίσεις, ε, δείχνει ότι όντως λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το θέμα του περιβάλλοντος. Ήταν μια νομοθεσία που εωθετήθηκε με τεράστια πλειοψηφία και πρέπει να το υπερασπιστούμε. Ο κύριος Κράμερ και μετά ο κύριος Σέγκχαουτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πριν από τρία χρόνια εγώ διαπραγματεύτηκα αυτή την οδηγία μαζί με τον εισηγητή και τους σκιώδες εισηγητές. Εγώ έχω κάπως διαφορετική εκτίμηση της κατάστασης σήμερα στην στιγμή όπου πολλοί εκτιμών στο Κοινοβούλιο είπαν ότι δεν θα πρέπει να υποτιμούμε το πρόβλημα που μπορεί να έχουμε με τρίτες χώρες. Δεν έχει νόημα να λέμε ότι ψηφίσαμε με συντριπτική πλειοψηφία τότε, το υπερψηφίσαμε μάλλον με συντριπτική πλειοψηφία. Γεγονό παραμένει ότι η διεθνής κατάσταση σήμερα είναι τελείως διαφορετική. Θα πρέπει πλέον να αναγνωρίσουμε πως υπάρχουν τρίτες χώρες που δεν θέλουν να συμμετέχουν και μάλιστα θέλουν να αντισταθούν στο σύστημα αυτό. Το ψήφισμα του ΙΚΑΟ, της ΙΚΑΟ πέρυσι θα έπρεπε να μας είχε προειδοποιήσει ότι υπήρχε πρόβλημα εδώ, ότι υπήρχε κίνδυνος και ότι έπρεπε να προβούμε σε δράση. Δεν μπορούμε απλώς να τα αφήνουμε λες και δεν τρέχει τίποτα. Δεν έχει νόημα όταν όλος ο κόσμος το βλέπει διαφορετικά. Και πιστεύω ότι η επιστολή της Χίλαρη Κλίντον προς την, επιστρο... προς την Επιτροπή ήταν ε, σαφής προειδοποίηση. Ε, μιλάμε για τη δημιουργία μιας ε, πολιτικής σύγκρουσης και όταν κοιτάω εδώ το καλάθι των πρωτοβουλειών πρέπει να πω ότι υπάρχει εδώ κίνδυνος πιθανότατα να υπάρξει πολιτική σύγκρουση. Και κλείνω, ε, θα πρέπει να προσέξουμε ε, η πολιτική ζαμιά αυτή η οποία έχει υποκληθεί ε, εδώ και πολύ καιρό να μην γίνει και οικονομική. Και δεν μιλάμε για το κόστος του συστήματος κύριε Λίζε, δεν είναι αυτό το σωστό επιχείρημα. Μιλάμε για παρέμβαση στα κυριαρχικά δικαιώματα άλλων χωρών. Έχετε ξεπεράσει το χρόνο σας, λέει ο Πρόεδρος. Και μετά τις διαπραγματεύσεις θα πρέπει να ε, ξεκινήσουμε νέα μέτρα. Ο Πας Άικχαουτ και η κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, πραγματικά με εντυπωσιάζει ο συνάδελφο Κράμερ, γιατί όταν συζητάμε για τα στοιχεία των επιβατών στη ΣΥΠΑ, δεν ακούω να λέει τίποτα για τι σχέσει μεταξύ Ένωση και ΗΠΑ. Είναι πρόθυμο να δώσει ε, τζάμπα τα στοιχεία αυτά. Και τώρα κάνουμε κάτι για το περιβάλλον με βάση την αρχή ο Ριπέρο πληρώνει, που είναι πολιτική αρχή και ακούμε αυτά τα μυστηρία επιχειρήματα. Γιατί τι συζητάμε τώρα εδώ, τι έγινε στη Μόσχα. Έκαναν και μια δήλωση με πολύ σαφείς δηλώσεις. Είναι ένα καλάθι γιατί δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν. Ο Καναδάς όταν ε, ε, δεν, μπορούσε, δεν συμφωνούσε στο Δελχή ήταν σύμφωνοι, μετά στη Μόσχα όχι πια. Τι κάνουν δηλαδή, ε, δοκιμάζουν ε, τους Ευρωπαίους νομοθέτες. Ε, θα χάσουμε την ψυχραιμία μας ή όχι. Ορισμένοι ναι, αλλά ξέρω ότι η κυρία Φώστερ θα μιλήσει αργότερα. Εκείνη αρχίζει και χάνει την ψυχραιμία της. Αλλά εγώ είμαι ευτυχής που το ΕΛΚ δεν χάνει την ψυχραιμία του. Η πράσινη πάντως σίγουρα όχι. Πού είναι η Άλντε λοιπόν, πού βρίσκεται η Άλντε. Άκουσα τον κύριο Κράμερ και πραγματικά ειλικρινά ελπίζω να μην μιλάει εξ ονόματος της ομάδας Άλντε. Γιατί τότε η αρχή ορυπαίνων πληρώνεις, ε, πληρώνει τη Άλντε, θα μείνει απλά στα λόγια. Η κυρία Φώστερ και κατόπιν η Λίντα Μακέβαν. Um, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Νομίζω πως ε, όλοι εδώ διαμαρτύρονται υπερβολικά. Έχουμε διαφορετικές απόψεις ε, για διάφορα θέματα. Γι' αυτό ε, υπάρχουν τα κοινοβούλια. Εγώ τυχάνει να συμφωνώ με τον κύριο Κράμερ. Δεν ξέρω αμφισβητώ το πόσο χρόνο έχουμε εδώ για αυτή τη σημαντική συζήτηση, γιατί υπάρχουν εδώ τεράστια δεκυβεύματα. Δεν είναι αρχή, το, το θέμα του κατά πόσο είναι καλό να υπάρχει το ETS ή όχι. Και είναι καλό που ακούμε να συζητάμε την ΙΚΑΟ η Κομισιόν, αλλά είναι κρίμα που δεν έγινε προηγούμενα, ότι, όπου υπήρξε προειδοποίηση που έλεγε ότι δεν μπορείς να φορολογήσεις τρίτες χώρες, ε, έξω εδαφικότητα. Κανείς δεν τα άκουσε τότε και τώρα είμαστε σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Ε, είμαστε σε μια θέση όπου έχουμε πρόβλημα με παραγγελίες για τους παραγωγούς εδώ στην Ευρώπη. Στην ε, κατασκευαστική εταιρεία έχουμε 8 δις ε, παραγγελίες που είναι υπό απειλή. Η απόφαση να μην ακούσουμε πριν από κάποια χρόνια και να μην συζητήσουμε σωστά με τις τρίτες χώρες ποιο ήταν ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε μας έχει θέσει σε μια ε, κατάσταση όπου όταν μιλάμε για εμπορικούς πολέμους εδώ έχουμε μια από τις πιο α, ε, συγκρουσιακές καταστάσεις που έχω ποτέ συναντήσει εδώ στο Κοινοβούλιο. Μόνο η Κομισιόν ε, θεώρησε ότι μπορούσε μάλλον με τη στάση της μπόρεσε να τους ε, συγκεντρώσει και να κάνει να συμμαχήσουν όλοι εναντίον μας. Ρώσοι, Κινέζοι, Ινδοί ε, και όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Δεν είναι διεθνή αυτή η συμφωνία. Τουλάχιστον θα έπρεπε να φτάσουμε σε μια διεθνή συμφωνία. Αλλά τώρα είναι θέμα ανταγωνισμού, Πρόεδρε. Γιατί τι λέμε, από την αρχή του, από την 1η Ιανουαρίου, υποτίθεται ότι όλοι πρέπει να συμμορφωθούν. Όλε οι ευρωπαϊκέ εταιρείε πρέπει να συμμορφωθούν. Αλλά αυτό που κάνουν είναι ότι οι τρίτε χώρε δεν θα συμμορφωθούν. Άρα είμαστε, έχουμε ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Είναι πραγματικά η κατάσταση χάλια. Μιλούν μαζί. Ο, η και ο πρόεδρος δεν καταλαβαίνουμε τι λένε. Η κυρία Μακάβανο. Εγώ υποστηρίζω, όπως και ο Ματία Γκρότα την Κομισιόν. Έχουμε κάνει αυτή την ε, συζήτηση. Έχουμε κάνει συζητήσεις, τζάκι, πριν, ε, με διάφορες χώρες πριν να νομοθετήσουμε. Το γεγονός ότι η ΚΑΟ λέει τώρα ότι κάτι θα κάνει είναι νίκη της Ένωσης. Εάν εμεί δεν είχαμε κάνει τίποτα, δεν θα είχαν κάνει τίποτα και αυτοί. Και αν καταλήξουμε σε καλά μέτρα, εντάξει, τα ξαναεξετάσουμε. Έχουμε μια νομοθεσία. Δεν υπάρχει καμιά πρόταση όμως επιτάπητο. ούτε και το Συμβούλιο δεν έχει κάνει πρόταση, γιατί το υποστήριξαν. Η Βρετανική κυβέρνηση στηρίζει αυτή την πρόταση της Κομισιόν. Το στηρίζει το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει πρόταση για απόσυρση αυτή τη νομοθεσία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε και να την εφαρμόσουμε αυτή τη νομοθεσία. Ευχαριστώ, Κρί Davis και μετά ο Τζο Λάινεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν τα κράτη-μέλη θέλουν να επιβάλλουν φορολογία στι, ε, στις αερομεταφορές, μπορούν να το κάνουν και όπως ο Πίτερ Λίζε είπε, ε, οι φόροι είναι ε, πολύ λιγότεροι από το, τα τέλη για το ETS. Αλλά έχουμε συμφωνήσει πάνω στο ETS, όλοι το γνωρίζουν. Τώρα αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση όπου οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο λένε ότι δεν μας αρέσει αυτό. Ε, και ο Πας ε, ε, λέει η Άλντε τι γνώμη έχει. Εγώ δεν ξέρω ποια είναι η θέση μου, η θέση μας, αλλά να μαντέψω με βάση αυτά που έχω ακούσει από τον Κίφερ Χόφστατ. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει απόφαση και ο υπόλοιπο κόσμος λέει ότι δεν μας αρέσει αυτό και δεν είμαστε διατεθειμένοι να το δεχτούμε, τότε ο Γκί τότε λέει ότι θα πάρει το μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέμε ότι ε, αυτό ισχύει για τα αεροπλάνα που χρησιμοποιούν τα δικά μας αεροδρόμια. Θέλουμε να στείλουμε ε, ένα σαφές μήνυμα προς την ε, Επιτροπή ότι στηρίζουμε τις προσπάθειές της, θέλουμε μια διεθνή συμφωνία, θέλουμε η ΚΑΟ να κινηθεί προς μια κατεύθυνση που να μπορούμε να δεχτούμε και δεν θα υποχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, Κριστέιβης. Ο Τζο Λάινεν και κατόπιν ο κύριος ε, Κερπράντη. Ναι, αυτή η μυστική συνάντηση στη Μόσχα σίγουρα ε, ε θέτει ε, σε αμφισβήτηση την αξιοπιστία της πολιτικής για το κλίμα αυτό είναι μια δοκιμή των ε, ομάδων ε, συμφερόντων, ε, των λόμπι, διότι θέλουν να δουν πόσο ισχυρή είναι η νομοθεσία για το κλίμα. Βρίσκω περίεργο αυτό που είπε ο συνάδελφος Κράμερ ότι το ETS αποτελεί ε, παρέμβαση στην, ε, στα κυριαρχικά δικαιώματα ε, άλλων χωρών. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Υπάρχουν τέλη προσγείωσης, υπάρχουν ένα σωρό άλλα τέλη στις αερομεταφορές. Γιατί ειδικά το ETS, το σύστημα εμπορίας εκπομπών, αποτελεί επέμβαση στα κυριαρχικά δικαιώματα και αυτό που ε, είπε η Ρωσία να μην επιτρέπει ε, τα αεροσκάφη να ε, πετούν πάνω από την Σιβηρία, αυτό είναι παρέμβαση και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά αυτή την απειλή. Δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποτύχει. Νομίζω ότι βρισκόμαστε καθοδόν προς μια επιτυχία. Δεν θέλουμε βέβαια εμπορικό πόλεμο. Εάν η ΚΑΟ μετακινηθεί και αν ο πρόεδρος ε, συγκεντρώσει ε, όλους ε, για να δημιουργηθεί ένα σύστημα που να μπορεί να εφαρμοστεί, τότε αυτό θα είναι καλό. Νομίζω ότι θα πρέπει να παραμείνουμε ψύχρεμοι. Ευχαριστούμε, Τζο Λάινεν. Δύο μιλητές έχω στον κατάλογο. Κερπράντι και Σάτου Χάση. Ευχαριστώ. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της πολιτικής για το κλίμα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε μόνο... Ε, δεν έχουμε ένα νέο πλαίσιο. Ε, και μάλιστα είναι και διασυνοριακός ο χαρακτήρας της α, ε, αεροπορίας, εξορισμού. Γι' αυτό και θέλουμε συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού. Προτείνω, προτιμώ μια διεθνή ε, λύσει σε επίπεδο Διεθνού Οργάνωση Πολιτική Αεροπορία. 20 χρόνια ήταν αναποτελεσματικέ οι Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σύστημα εμπορία εκπομπών ω μέσο πίεση. Και συμφωνώ με τον ε, κ. Ακχάουτ για τι αδυναμίε τη ομάδα τη Μόσχα ε, και είναι και πολύ ατερόκλητο αυτό ο συνασπισμό. Ακόμη και η Λευκορωσία, που είναι από τι πιο απομονωμένε χώρε του κόσμου, συμμετέχει σε αυτή τη συμμαχία. Και μάλιστα έδιωξαν τον Ευρωπαίο πρέσβη ε, την περασμένη εβδομάδα. Δεν νομίζω ότι κανεί θέλει να ανοίξει σε συμμαχία τέτοιων χωρών. Πάντω, η στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι εμένοντα το ETS βλέπει να γίνονται κάποιε κινήσει υπέρ μια παγκόσμια συμφωνία και στην Παγκόσμια Οργάνωση Πολιτική Αεροπορία. Οπότε, αν εμεί τώρα υπαναχωρήσουμε, θα κάνουμε λάθος, θα πρέπει να συνεχίσουμε τις πιέσεις. Εγώ πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να επιτύχουμε παγκόσμια λύση στα πλαίσια της ΑΕΚΑΟ που θα την προσυπογράψουν όλοι και ο μεγάλος κερδισμένος αυτής της ιστορίας είναι τελικά το κλίμα. Ευχαριστώ η κυρία Σάτου Χάση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Κερμπράντη και συμφωνώ πλήρως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει όλοι καταλάβουμε ότι ο νόμος είναι νόμος. Ο νόμος αυτός ε, ε το... οριστικοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2008, ενώ η αρχική πρόταση είχε υποβληθεί το 2006 και κανένας ε, δεν εφηνεδιάστηκε. Το 1997 στο Κιώτο ανέλαβε η ΚΑΟ την ε, υποχρέωση να υποβάλει μια πρόταση διεθνώς και τελικά δεν έκανε τίποτα. Μια τρύπα μες στο νερό αδράνησε. Ε, ερμήνευσε την κατάσταση ως ε, ο καθένας κάνει ό,τι του κατέβει στην πολιτική του κλίματος. Ε. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί αυτή η κατάσταση, αυτό το ξέφραγο αμπέλι να συνεχιστεί επαόριστο. Ο νόμος είναι νόμος και εμείς έχουμε δικαίωμα να υποβάλουμε ρυθμίσεις και να θεσπίζουμε νομοθετικά μέτρα εντός επικράτειάς μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έτσι ολοκληρώσαμε το κατάλογο των ομιλητών. Να δώσω το λόγο στην Κομισιόν, στον ε, Γενικό Διευθυντή ε, για το κλίμα. Αν ε, μπορείτε, παρακαλώ, περιοριστείτε στα πέντε λεπτά, διότι έχουμε ένα ακόμα σημαντικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Σας παρακαλώ, σύντομα. Well, thank you very much. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι συναπτική χωρίς όμως να παραλείπω τα βασικά στοιχεία της συζήτησης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής σας, γιατί σε μεγάλο βαθμό υποστηρίξατε την κοινοτική νομοθεσία, που είναι ουσιαστικά νομοθεσία για, την, για το περιορισμό των κλιματικών αλλαγών. Και όπως ε, είπαν πολλοί ευρωβουλευτές, είναι θέμα αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κλιματικές αλλαγές ε, αποτελούν αντικείμενο μιας ε, από τις σημαντικότερες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και περιλαμβάνονται στις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες μας. Έχουμε κοινοτική νομοθεσία που από κοινού θέσπισαν το Κοινοβούλιο με το, Ευρωπαϊκό, με το, με το Συμβούλιο. Έχουμε λοιπόν σημαντική μόχλευση για να προωθήσουμε τη συζήτηση παγκοσμίω στο επίπεδο της ε, Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας. Τώρα θα ήθελα να ασχοληθώ με μερικά επιμέρους ζητήματα που αναφέρθηκαν. Καταρχήν, σε σχέση με τη διάσκεψη της Μόσχας. Είπατε κι εσείς ότι η διάσκεψη κορυφής της Μόσχας Ήταν ένα φόρουμ για πολλά μέλη της ΑΙΚΑΟ που συμφώνησαν να συνεργαστούν και σε επίπεδο ΑΙΚΑΟ και κατέθεσαν και μία σειρά προτάσεων για μέτρα που μπορούν να εξεταστούν. Πάντως, αν δούμε το σχέδιο δήλωσης της διάσκεψης αυτής και την τελική δήλωση, που υπευλήθηκε διαπιστώνουμε ότι τελικά το αποτέλεσμα έδειξε μια διαραγή του μετόπου σε ό,τι αφορά τις απαραίτητες δράσεις. Πάντως, αυτό που είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι ότι οι χώρες που συμμετείχαν και στη Μόσχα συμφωνούν υπέρ μιας συζήτησης στην ΕΚΑΟ. Όπως σας είπα, η ελαστικότητά μας αφορούν τις ερχόμενες πτήσεις. Δεν λέμε σε κανέναν σε καμία αερογραμμή του κόσμου ότι δεν μας ενδιαφέρουν οι δράσεις που θα αναλάβουν εκείνοι. Μας ενδιαφέρουν και οι δράσεις των υπόλοιπων χωρών. Και έχουμε και ελαστικές ειρήτερε στην νομοθεσία μας, προκειμένου να λάβουμε υπόψη και δράσεις που αναλαμβάνουν και άλλες χώρες για να μειώσουν τις εκπομπές αερίων ε, του θερμοκηπίου της πολιτικής αεροπορίας. Πάντως νομίζω ότι όντως το σύστημα εμπορίας εκπομπών της Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταλητικό ρόλο και παγκοσμίω. Γνωρίζω ότι δεν συμφωνείτε όλοι με την άποψη αυτή, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της ΑΙΚΑΟ. Γιατί κατά τη γνώμη μας αυτό είναι το κατάλληλο φόρουμ για τη συζήτηση. Άλλωστε, χρειάστηκε να περιμένουμε 15 χρόνια για παγκόσμια δράση προκειμένου να κινητοποιηθούμε εμείς και να λάβουμε τα δικά μας μέτρα. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθούμε να πιστεύουμε έθερμα ε, ότι ο κατάλληλος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, με παγκοσμίως ε, ε, αποδεκτά μέτρα. Κύριε Πρόεδρε, Θα ήθελα να απαντήσω σε όσους ρώτησαν ποιο θα είναι το κόστος αυτού του μέτρου. Δεν νομίζω ότι η συζήτηση αυτή αφορά τόσο το οικονομικό κόστος. Αν δείτε το κόστος για την αεροπορία, βλέπουμε ότι παρά το σύστημα εμπορία εκπομπών δεν έχουν ακριβήνει πολύ τα αεροπορικά εισιτήρια. Και αν δείτε τους υπολογισμούς των ερευνητών, των μελετητών, θα διαπιστώσετε ότι ε, ένα αεροπορικό στήριο μπορεί να αυξηθεί λιγότερο από 2 ευρώ για τις μεγάλες πτήσεις. Δεν είναι θέμα κόστους λοιπόν, είναι περισσότερο θέμα πολιτικής και αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ανέκαθεν αξιόπιστη και ήταν ανέκαθεν πρόθυμη ε, για συνεργασία σε πολυ... πολυμερές επίπεδο και χαιρόμαστε για την υποστήριξή σας. Γιατί πιστεύουμε ότι διάλογος θα πρέπει να γίνει διεθνώς με τους υπόλοιπους εταίρους σε πολυμερές επίπεδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις εξηγήσεις που μας δώσατε και ε, για την ε, θερμή υποστήριξή σας ε, για αυτό το νομοθέτημα. Μπορώ να σας πω ότι η πλειοψηφία της ε, Επιτροπής μας ε, θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε ε, να περάσουμε το τεστ για αυτό το θέμα. Περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης. Πρόκειται για το 19. Κλινικές δοκιμές στις χώρες με χαμηλό εισόδημα. Το ζήτησε αυτό ο συνάδελφος ε, Πέτερ Λίζε, του δίνω κατευθείαν το λόγο. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ναι, τους τελευταίους μήνες ήρθαν σε επαφή μαζί μου πολλοί εμπειρογνώμονες ε, για το θέμα αυτό και είχαμε στο Στρασβούργο μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ άλλων με έναν Ινδό καθηγητή ο οποίος μας έδειξε πως για παράδειγμα στην Ινδία αλλά και σε άλλες χώρες με χαμηλό εισόδημα πραγματοποιούνται κλινικές δοκιμές και δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι φάρμακα φάρμακα τα οποία διατίθεται στην αγορά της Ευρώπης εν μέρη ε, έχουν ε, ε, δοκιμαστεί σε τρίτες χώρες και παρότι ε, ε, λένε τα πρότυπα τα οποία έχουμε θέσει, ε, η νομοθεσία που έχουμε θεσπίσει λέει ότι πρέπει να τηρούνται τα πρότυπα. ακούμε ότι δεν τηρούνται τα πρότυπα ασφαλείας, άνθρωποι πεθαίνουν και αυτό βέβαια μπορεί να έχει επιπτώσεις και σε ζωές ανθρώπων στην Ευρώπη διότι αν δεν τηρούνται τα πρότυπα, αν δεν πληρούνται τα πρότυπα τότε μπορεί να μην είναι ασφαλή τα φάρμακα. Ε, η ΕΜΑ και η ΕΟΦ, δηλαδή και η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν εντοπίσει το πρόβλημα. Χρειαζόμαστε όμως μεγάλη πολιτική υποστήριξη για το θέμα αυτό. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε την ε, νομοθεσία, διότι η νομοθεσία λέει ότι τα πρότυπα που ισχύουν στην Ευρώπη για τις κλινικές δοκιμές θα πρέπει να ε, τηρούνται για να ε, εγκριθεί ένα φάρμακο στην Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμόζεται καλύτερη η νομοθεσία. Θα παρακολουθήσω λοιπόν την Κομισιόν και την, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων να μας πούν τι έχουν κάνει ήδη, τι πρέπει να γίνει, πώς χρειάζεστε την η υποστήριξη το, του Κοινοβουλίου. Αν ε, μου πούν όμως ότι αρκούν αυτά που ήδη γίνονται, αυτό δεν μου αρκεί ως απάντηση. Ε, ευχαριστώ πολύ, Επιτελίζε. Θα ήθελα καταρχήν να σας πω ότι ε, έχουμε εδώ μια ομάδα τηλεοπτική από το κανάλι VDR της Γερμανίας. να δώσω τον λόγο στην Κομισιόν για πέντε λεπτά, ώστε και η Έμα να μπορέσει να πάρει το λόγο ο ΕΟΦ δηλαδή, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και να μπορέσουμε να έχουμε συζήτηση. Παρακαλώ. Ich hoffe, die technischen Schwierigkeiten sind... Ελπίζω να έχουν ξεπεραστεί οι τεχνικές δυσκολίες. Εκ μέρους της Κομισιόν είναι παρόν. Ο κύριος Σέρο, παρακαλώ. Thank you, Mr. Chairman. Uh, well, uh, first of all, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ευχαριστώ τον κύριο Λίζα για την πρόσκληση και για το ότι τοποθέτησε αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη. Εγώ είμαι νεοφερμένο εδώ, οπότε ελπίζω πως θα κάνετε υπομονή μαζί μου. Καταρχήν να πούμε τι είναι μια κλινική δοκιμή είναι η δοκιμή ενός φαρμάκου επί ανθρώπινων όντων. Ένα τέτοιο φάρμακο μπορεί να είναι ήδη εγκεκριμένο ή όχι. Δεν είναι υψηλοκίνδυνο κινδύνου εγχείρημα. Σημαίνει ωφέλη για την κοινωνία για... και πιθανότατα και για τον ασθενή, δηλαδή το υποκείμενο της δοκιμής της κλινικής δοκιμής. Το υποκείμενο αυτά συχνά για ειδικά θέματα ιδιωτικού τομείς ιατρική θέλουν να συμμετέχουν στις κλινικές δοκιμές. Αρχικά στην Ένωση έχουμε μια ανησυχητική εικόνα. Υπάρχει μείωση των κλινικών δοκιμών. Τα τελευταία χρόνια, από το 2007 μέχρι και το 2010, χάσαμε 15% των εφαρμοσμένων κλινικών δοκιμών στην Ένωση και το ίδιο πτωτική στάση φαίνεται να υπάρχει και για το 2011. η οδηγία του 2001 για τις κλινικές δοκιμές είναι ίσως η πιο αυτή η νομοθεσία η οποία επικρίθηκε περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όσον αφορά την πολιτική της, ε, για την υγεία. Συχνά υπόθηκε πως ε, σε αυτήν οφείλεται η μείωση των κλινικών δοκιμών. Κατά τη γνώμη μας δεν είναι μόνο το μόνο αίτιο, αλλά είναι ένα από τα αίτια. Προσπαθούμε τώρα αυτό να το αλλάξουμε και να υποβάλουμε μια πρόταση στα μέση του 2012. Αυτό δεν είναι το κεντρικό θέμα της συζήτησης, οπότε δεν θα σας κουράσω με τις λεπτομέρειες του τι σκοπεύουμε να κάνουμε και θα εστιάσω στο θέμα της σημερινής συζήτησης. Είδαμε λοιπόν ότι υπάρχει μείωση όσον αφορά την ελκυστικότητα των κλινικών δοκιμών στην Ευρώπη και είναι σημαντικό να μείνει κανείς ελκυστικός. Είναι μια παγκόσμια ε, υπόθεση σε, μια παγκόσμια χώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, είναι πια ένα μικρό σημείο σε έναν μεγάλο χάρτη. Η εικόνα που έχετε μπροστά σας δείχνει την τοποθεσία ε, των ασθενών ε, το, από το 2007 μέχρι το 2009 σε τρίτες χώρες για ε, κλινικές δοκιμές κλειδιά. Εν ολίγης, το 1 τρίτο των κλινικών δοκιμών γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 1 τρίτο στην Βόρεια Αμερική και το άλλο τρίτο στην υπόλοιπο κόσμο. Κυρίως στις αναδυόμενες χώρες, εκεί, δηλαδή οικονομίες εκτός της Αφρικής. Υπάρχει ένα σύνολο κανόνων, και, αλλά πιστεύουμε ότι η απόπειρα για παγκοσμιοποίηση των κανόνων δεν είναι αρνητική. Υπάρχουν κάποιες διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές που ασχολούνται με την ηθική ε, και τα θέματα ασφάλειας, ιδιαίτερα οι καλές κλινικές πρακτικές του ICH αλλά και ε, σε επίπεδο ΟΗΕ και Συμβουλίου της Ευρώπης υπάρχουν σχετικές συστάσεις. Υπάρχουν δύο νομοθεσίες. Η μία είναι η οδηγία για τις κλινικές δοκιμές που λέει πώς θα πρέπει να γίνονται αυτές και το άλλο είναι ο κοινοτικό κώδικα ε, φαρμάκων που λέει, ότι ποιες, που λέει ποιες θα πρέπει να είναι οι κλινικές δοκιμές στις οποίες θα πρέπει να περάσει ένα φάρμακο για να αδειοδοτηθεί. Υπάρχουν ανησυχίες για τις τρίτες χώρες, για το κατά πόσο αυτές ε, ζητούν αυτή την ε, αδειοδότηση, αλλά υπάρχουν ε, περιορισμοί όσον αφορά τη δικαιοδοσία και τις αρμοδιότητες της. Όσον αφορά τις κλινικές δοκιμές σε τρίτες χώρες, ο κοινοτικός κώδικας για τα φάρμακα λέει ότι τα στοιχεία κλινικών δοκιμών που έχουν ε, προκύψει στην Ένωση και τα δεδομένα ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ισχύουν ε, εφόσον έχουν εκδοθεί με αντίστοιχα στάνταρ. αυτό ισχύει, αλλά δεν πιστεύουμε ότι μπορεί κάτι τέτοιο να γίνει πιο λειτουργικό μέσω αλλαγή τη νομοθεσία. Είναι περισσότερο ένα θέμα εφαρμογή της νομοθεσίας που υπάρχει, που ισχύει. Δεν θέλουμε να είναι πιο περιοριστικές οι κλινικές δοκιμές, ώστε περισσότερες κλινικές δοκιμές να γίνονται εκτός Ένωση. Θέλουμε να πετύχουμε καλύτερη παγκόσμια ευθυγράμμιση τη νομοθεσία, καλύτερη παγκόσμια συνεργασία στην δημιουργία δυνατοτήτων. Πολλά συμβαίνουν και αυτά αφορούν την ε, επιβολή και όχι νέους νόμους, ε, ε, επιθεωρήσεις και διαφάνεια. Σύντομα, σε 20 δευτερόλεπτα να σας πω ότι η παγκοσμιοποίηση στην ε, κλινική έρευνα υπάρχει, δεν είναι αρνητική. Εδώ δεν θέλουμε να αλλάξουμε τους κανόνες, αλλά να επιβάλλουμε, να επιβάλλουμε και να επιβάλλουμε τους υπάρχοντες. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας και θα ακούσουμε τώρα την παρουσίαση του εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, του κυρίου Φέργκουσον. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας παρακαλώ, αν μπορείτε, να περιοριστείτε και εσείς τα πέντε λεπτά, ώστε να μπορέσουν οι συνάδελφοι να θέσουν συγκροματικές ερωτήσεις. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τον δακτωρα Λίζε που περιέλαβε αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη και μας δίνει την ευκαιρία να λάβουμε το λόγο εδώ σήμερα. Ε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ΕΟΦ, προσπαθεί να εντοπίσει ε, την ε, προέλευση ε, φαρμάκων που χρησιμοποιούνται σε κλινικές δοκιμές και όπως ακούσαμε και προηγουμένως έχουμε τα περισσότερα φάρμακα αυτά από την Ευρώπη, από τη Βόρεια Αφρική και ελάχιστα από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου όπως βλέπετε στη διαφάνεια. Πάντως αυτές οι κλινικές δοκιμές αφορούν τρία τέταρτα των ασθενών 57.000 κλινικές δοκιμές, μερικές φορές για 2-3 κλινικές δοκιμές για το ίδιο φάρμακο. Και από 90 χώρες έχουμε δώσει 400, έχουμε λάβει 400 αιτήσει για εμπορία και είχαμε 215 ελέγχους που εγκαινιάσαμε εμείς στον ΕΟΦ. Και μάλιστα ε, γίνονται από επιθεωρητές των κρατών μελών. Δεν έχουμε εμεί σχετική νομική αρμοδιότητα και επίσης πολλές ε, επιθεωρήσεις και έλεγχοι γίνονται εντός της Ευρώπης. Γιατί είναι σημαντικό και εμείς στην Ευρώπη να κρατήσουμε τάξη στον οίκο μας. Βλέπετε στη διαφάνεια, δεν, είναι εύκολο να τη διαβάσετε, πάντως βλέπετε πόσες κλινικές ε, δοκιμές γίνονται στις διάφορες αιτήσει για εμπορία εκτός της Ευρώπης, κυρίως στη Βόρεια Αμερική και βλέπετε την κατανομή αναχώρα. Και αυτό είδατε και στη διαφάνεια του κυρίου Σόρο. Μετά τον, τις ΗΠΑ και τον Καναδά έχουμε τη Ρωσία, τη Βραζιλία, την Νότια Αφρική, την Αργεντινή, την Ινδία, το Μεξικό. Από αυτές τις χώρες περιμένετε να έχουν γίνει ήδη κλινικές δοκιμές. Φέτος στην Ιδία Κίνα έχουμε πολύ μεγαλύτερη δραστηριότητα, πολύ, περισσότερα, πολύ περισσότερες περιπτώσεις από αυτές που βλέπετε. Τώρα, τώρα βλέπετε την αύξηση των ελέγχων από το 2000 ε, μέχρι το 2010, αριστερά το 2000, ε, ε, δεξιά το 2010 και βλέπετε την κατανομή των ελέγχων στην Ευρώπη και τις Ηνωμένε Πολιτείες, ιδιαίτερα από το 2007, όπου εφαρμόσαμε μια νέα αναθεωρημένη πολιτική επιθεωρήσεων και ελέγχων στις διάφορες περιοχές του κόσμου. Και βλέπετε εδώ τις χώρες στις οποίες έχουν γίνει σχετικές ε, επιθεωρήσεις και έλεγχοι από τις διάφορες υπήρους. Σε ό,τι αφορά ε, την πραγωγή του όρου της ισοδυναμίας των κλινικών δοκιμών, έχουμε αυτό το έγγραφο για τις κλινικές δοκιμές ε, για τη θέση σε εμπορία και την αδειοδότηση. Αυτό έγινε μετά από διεθνείς διαβουλεύσεις με ρυθμιστικές αρχές, ε, χορηγούς ε, και άλλους ενδιαφερόμενους. Και το έγγραφο εντοπίζεται σε τέσσερις τομείς. Διεθνή συνεργασία, έμπρακτη εφαρμογή των διοντολογικών προδιαγραφών, ε, φυσικά σε πρακτικό επίπεδο, τα βήματα που θα πρέπει να γίνουν πριν την έναρξη της κλινικής ε, δοκιμής ε, σε ό,τι αφορά την παροχή συμβουλών, τις κατευθυντήρες γραμμές, καλύτερα να βελτιώνουμε σε προκατακτικό επίπεδο από το να επικρίνουμε αργότερα και φυσικά εξακρίβωση της συμμόρφωσης. Αυτό γίνονται από τις διάφορες επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν γιατροί, εκπρόσωποι των ιατρικών υπηρεσιών, καταναλωτών κτλ. Τα βασικά σημεία δεν υπάρχουν νομικά κριτήρια και απαιτήσει. Φυσικά έχουμε το σαφές μήνυμα ε, των δεντολογικών προδιαγραφών, εφαρμογή δραστηριών μέτρων προκαταρκτικά, ιδιαίτερα με ε, παροχή συμβουλών σε χορηγούς, σε κρατημέλη ή διαλογή ε, και επίσης περίπτωση παροχής τεχνογνωσίας σε δύσκολες περιπτώσεις γιατί τα συμπεράσματα δεν είναι εύκολα και επίτεση της διαφάνειας πολύ σημαντικό και φυσικά το θέμα της προέλευσης των ασθενών και ιδιαίτερα ευάλωτοι ασθενείς. Εδώ έχουμε κάποιες λεπτομέρειες από τις έκθεσεις του Διεθνούς Σεμινάριου που έγινε ενίσχυση και πάλι έχουμε της διεθνούς συνεργασίας ε, υπό την αιγίδα ε, διαφορών συμφωνιών και διμερών συζητήσεων στις οποίες συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με Κίνα, Ινδία, Ρωσία, με την Παγκοσμία Οργάνωση Υγείας προκειμένου να διαμορφωθεί ένα παγκόσμιο πλαίσιο. Έχουμε επιθεωρητές της ΕΠΗ από πολλές χώρες, επιτροπές συνδεδολογίας, πολλές πρωτοβουλίες και τα επόμενα βήματα η δημοσίευση του αναθεωρημένου εγγράφου και συνεχίζουμε φυσικά τις, ε, την επικαιροποίηση προκειμένου να ενημερώσουμε καλύτερα και να συμπληρώσουμε τον τοσχέ για τις κλινικές δοκιμές, ε, να δώσουμε τεχνογνωσία στις χώρες με χαμηλό εισόδημα και να συνεχίσουμε φυσικά την ε, σύσφυξη της διεθνούς συνεργασίας. Φυσικά θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πρόσφορο κλίμα και να έχουμε την εμπιστοσύνη ότι όλες οι χώρες εξυπηρετούν τους ασθενείς και φροντίζουν για το καλό τους. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας, η Άννα Ρόσπαχ, η Λίντα Μακέβαν και ο Πέτερ Λίζε. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ σήμερα ε, για να συζητήσετε μαζί μας αυτό το σοβαρό θέμα. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Τι συγκεκριμένα βήματα θα ληφθούν ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν παραβιάζονται οι κατευθυντήριες γραμμές στο μέλλον. Θα θέλαμε να ξέρουμε ποιο ήταν το πρόβλημα μέχρι τώρα, διότι λέτε ότι δεν χρειάζεται νέα νομοθεσία. Θα χρησιμοποιήσετε το, παρόν, το υπάρχον πλαίσιο. Τότε γιατί υπήρξαν προβλήματα, πού αποτύχαμε. Επίσης θα θέλαμε να γνωρίζουμε εάν η αίμα έχει επισκόπηση των ε, εταιριών και των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από τις ε, δοκιμές αυτές. Μιλάμε για πολλές επιχειρήσεις ή για λίγο και πόσες από τις επιχειρήσεις αυτές είναι ευρωπαϊκές. Ε, μιλάμε για κατεξακολούθηση παραβάτες και τέλος θα ήθελα να ξέρω τι τύπου κυρώσεις έχουν εφαρμοστεί, ε, έχουν επιληθεί στις επιχειρήσεις αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η Λίντα Μακέβαν. Ακούσαμε πολλές πληροφορίες τα τελευταία δέκα λεπτά. Είναι δύσκολο να αφομοιώσει κανείς όλες τις πληροφορίες αυτές. Ε, ας ε, μην κάνουμε σαν να μην υπάρχουν πολύ σοβαρέ ε, κατηγορίε. Εσεί μιλήσατε με κάποιον ε, από την Ινδία. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτέ τι περιπτώσει, αν ακουστούν σοβαρέ κατηγορίε, οι επιχειρήσει που ζητάνε αδειοδότηση από, την, τον ΕΟΦ για κάποια φάρμακα. Τι κάνει ο ΕΟΦ, πώς, τι κάνετε κατά τη διάρκεια της ε, διαδικασίας αδειοδότησης και όσον αφορά την βάση δεδομένων για τις κλινικές δοκιμές. Ε, πέρσι επιτέλους ε, μπήκε στο διαδίκτυο Έγινε επιγραμμική. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε. Από ό,τι καταλαβαίνω, ε, περιέχει τι ε, κλινικέ δοκιμέ που γίνονται εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δείχνει και κλινικέ δοκιμέ εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αρχίσει να δείχνει τέτοιε σε περίπτωση αρνητική από ό,τι κατάλαβα μιλάμε για παιδιατρικές κλινικές δοκιμές μόνο. Ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε ε, φαίνονται και τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών ε, στην επιγραμμική βάση δεδομένων. Ε, μου είπατε ότι δεν χρειάζεται να αλλάξει τίποτα, αλλά δεν, μήπως χρειαζόμαστε του ιδίου τύπου διαφάνεια με τις ε, Ηνωμένε Πολιτείε. Μήπως χρειάζεται να τροποποιήσουμε την οδηγία. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα ο Πέτερ Λίζε. Ε, πολύ σύντομα Καταλαβαίνω ότι δεν ε, χρειαζόμαστε ε, πιο αυστηρή νομοθεσία εντό Ευρώπη. Θα πρέπει να φροντίσουμε να, ε, όταν δίδονται άδεια σε φάρμακα εντό τη Ευρώπη, να φροντίζουμε να έχουν τηρηθεί τα πρότυπα και εκτό Ευρώπη. Ε, όσον αφορά τον κανόνα αντιστοιχίας θα ήθελα να μου πείτε και ε, θα ήθελα επίσης ε, να ξέρω όπως και η Λίντα Μακέβαν ε, να γνωρίζω πώς αντιδράτε σε περίπτωση κατηγοριών και ο κύριος Σουίνι ήταν στο Στρασβούργο και άκουσε την ομιλία του καθηγητή Γεράνη από την Ινδία και θα ήθελα και, και επίσης αν συνεργάσει τον κύριο Ζόρο εκεί θα ήθελα λοιπόν να ξέρω τι κάνει ο ΕΟΦ στι περιπτώσει αυτέ όταν υπάρχουν τόσο σοβαρέ κατηγορίε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι στην Ινδία, χωρίς, δεν έχουν λάβει αποζημίωση, δεν ε, τηρήθηκαν οι κανόνες. Ποιες είναι οι συνέπειες από τέτοιες ε, αναφορές. Ευχαριστώ πολύ, Πετερλίζε. Να δώσω τον λόγο πρώτα στον κύριο Σόρο και κατόπιν στον κύριο Σουίνι. Παρακαλώ. Να απαντήσει σε ερωτήσεις. Okay, very briefly. Uh, I did not exactly say the new... Ναι, σύντομα. Δεν είπα ακριβώ πω δεν χρειάζεται μια νέα νομοθεσία. Θα ήταν αυτό αντίφαση. Κάνουμε νέα νομοθεσία. Αυτό που είπα ωστόσο είναι ότι το να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, μάλλον τους όρους για τις κλινικές δοκιμές και να τους κάνουμε πιο αυστηρούς δεν είναι η λύση στην Ευρώπη. Και Κατά συνέπεια αυτό επηρεάζει και τους πίνακες επιδόσεων που χρησιμοποιούμε για τις κλινικές δοκιμές εκτός Ευρώπης. Το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα είναι να είναι πιο διαφανείς οι κλινικές δοκιμές και άρα και αλλού να είμαστε πιο διαφανείς. Να ξέρουμε τι κλινικές δοκιμές γίνονται και πώς και πού. Τα αιτήματα για έγκριση φαρμάκων που βασίζονται κλινικές, σε κλινικές δοκιμές εκτός Ένωσης να είναι και αυτά πιο ε, σαφή. Βασικά αυτό είπα. Κυρώσεις. Θα πείσω το λόγο στον Φέργου Σφίνη. Αν σαφές ότι όταν γίνει ένα αίτημα ε, για διοδότηση με βάση κλινικές δοκιμές που δεν πληρούν τις ε, προδιαγραφές δεν θα ενεκρινόταν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τσόρο. Και τώρα κύριε Σφίνη. Σας ευχαριστώ για τις διάφορες ερωτήσεις. Θα πρέπει να επανέλθουμε καταρχήν στο θέμα του νομικού πλαισίου αυτό το οποίο έχει φτιάξει η ΜΑ είναι το τι μπορούμε να κάνουμε μέσα στο ισχύον πλαίσιο. Γιατί είναι σημαντικό να σημειωθεί νέα πρόοδος εντός αυτού του πλαίσιου, γιατί θα έπαιρνε χρόνο αν η νομοθεσία. Πιστεύω ότι ένα θέμα κλειδί είναι το θέμα των πόρων. Βασιζόμαστε στις πόρους της επιθεώρησης και εκεί πρέπει να επαληθευτεί κατά πόσο υπάρχει συμμόρφωση με τους κανόνες εντός της Ευρώπης αλλά και τις μελέτες που γίνονται εκτός Ευρώπης. Αλλά όπως μπορείτε να δείτε από τα νούμερα τα οποία σας έδειξα, είναι αδύνατο να επισκεφθεί κανείς όλα αυτά τα μέρη, ε, ούτε ακόμα και ένα μικρό ποσοστό και γι' αυτό πρέπει να συνεργαστούμε με τους ε, νομοθέτες εκεί όπου γίνονται οι δοκιμές αυτές, ώστε να βελτιώσουμε τις ικανότητές τους για την αποτελεσματικότητα του δικού του συστήματος επιθεώρησης, καθώς και να εξετάσουμε ποιο είναι το σύστημα ηθικής που επικρατεί. Τώρα συνήθως ξέρουμε την εταιρεία και την, το ερευνητικό ίδρυμα που έχει κάνει τις δοκιμές. Αυτά συμπεριλαμβάνονται στα ντοσιέ που λαμβάνουμε και ε, γενικά η διεξαγωγή δοκιμών ε, σε αυτές τις χώρες εκτός Ένωσης και Βόρειας Αμερικής ε, γίνονται όλο ένα και περισσότερο στις χώρες εκτός Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής όλο ένα και περισσότερο γίνονται οι δοκιμές σε ολόκληρο τον κόσμο για να μπορούν να έχουν αρκετά μεγάλο δείγμα. Φυσικά οι δοκιμές εκτός ε, ε, Ένωση είναι εκτός αρμοδιότητας τόσο των κατανομελών όσο και των ευρωπαϊκών ε, θεσμών. Τι μπορούμε να κάνουμε εκτός από το να απαγορέψουμε την κυκλοφορία του, εν λόγω φαρμάκου. Είναι σημαντικό μέσο, αλλά χρειάζεται αυτό το μέστρο, αλλά σημαίνει ότι έτσι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση οι ασθενεί στην Ευρώπη αλλά και σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες που περιμένουν τη δική μας έγκριση για να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα αυτά. Γι' αυτό και προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις εκθέσεις μας, να δούμε πού έχουν γίνει κάθε φορά οι δοκιμές, από πού προέρχονταν οι ασθενείς, κατά πόσο ήταν ευάλωτοι ή όχι, ποια ήταν τα βήματα που στα οποία προέβησαν οι εταιρείε και εμείς, ώστε να εξασφαλίσουν την προστασία των ασθενών και ούτω καθεξής. Και έτσι μπορούμε να εκθέσουμε και να χρησιμοποιήσουμε το, το φάρμακο. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε αρνηθεί την κυκλοφορία φαρμάκων και οι κλινικές δοκιμές κάποιες φορές συνέβαλαν. Αν και η μη συμμόρφωση κατά την γνώμη μας δεν είναι γεωγραφικό ζήτημα, είναι, οφείλεται στο κατά πόσο οι κλινικές δοκιμές έχουν γίνει σωστά και όταν αποτυγχάνουν, αποτυγχάνουν και εδώ και στη Βόρεια αλλά και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και μάλιστα οι δοκιμές που γίνονται σε αναπτυσσόμενες χώρες γίνονται με μεγαλύτερη προσοχή από ό,τι στην Ευρώπη. Έχει υπάρξει μεγάλη επέκταση των δοκιμών, κλινικών δοκιμών στις αναπτυσσόμενες χώρες και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να εφαρμόζουμε αυτές τις διάφορες πρακτικές ε, διαδικασίες που σας περιέγραψα, ώστε να παραμένουμε σε παγρύπνηση, γιατί ενώ μπορεί να μην έχουμε δει σημαντικές παραβιάσεις στις συγκεκριμένες δοκιμές που εμείς λάβαμε ή που ελέγξαμε, ε, θα μπορούσε κανείς να πει ότι καθώς πολλοί αρχίζουν και μπαίνουν στο παιχνίδι, ε, πιέζονται πολύ ευάλωτα και νέα νομοθετικά συστήματα. Οπότε μπορεί όντω να προκύψουν προβλήματα. Γνωρίζουμε τις διάφορες εκθέσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις έχουν γίνει δοκιμές από εταιρείε για προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ευρώπη, αλλά οι συγκεκριμένε δοκιμέ οι οποίες επικρίθηκαν δεν έχουν αποτελέσει τη βάση για αιτήματα αδειοδότηση εδώ στην Ευρώπη. Έχω συζητήσει και με τον εξάρτητο συντάκτη έκθεσης ε, μεταξύ άλλων. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, πόρους για να αυξηθούν οι δυνατότητες αλλά και για να αυξηθούν οι επιθεωρήσεις για τη βάση δεδομένων δουλεύουμε με βάση το σύστημα που, υπά, που, ισχύει. Ενημερώνουμε για τις κλινικές δοκιμές που γίνονται σε ένα ή περισσότερο μέρη στην Ευρώπη και για τις παιδιατρικές δοκιμές ε, και εκτός Ευρώπης έχουμε στοιχεία. Για τις υπόλοιπες δοκιμές δεν μπορούμε να τις ε, ε, καταγράψουμε. Οι βάσεις μας συμπεριλαμβάνουν, συμπεριλαμβάνουν στοιχεία και από δοκιμές σε ad hoc πληθυσμούς. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ σημαντική η συζήτηση αυτή. Δυστυχώς ε, δεν είχαμε πολύ χρόνο για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Ε, θα συνεχίσουμε πάντως ε, τη συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό. Σας εύχομαι επιτυχία στη συνέχεια των εργασιών. Εύχομαι καλό μεσημέρι στους συναδέρφους ε, και θα τα ξαναπούμε στις 3 η ώρα. με το θέμα των, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Τηλεπικοινωνιών.